Colleagues, I, uh, I think... Συνάδελφοι, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Είναι 9.36. Πριν ξεκινήσουμε κανονικά, θα σας παρακαλέσω να φορέσετε τα ακουστικά σας και να ακούσετε ένα μήνυμα από τους διερμηνείς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 το εργαστήριο για τις ε, εξαγωγές όπλων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ως πρώτο θέμα θα εξετάσουμε αυτό το θέμα στην μέσα Διαταξή σήμερα. Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα αυτό ούτως ή άλλως έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας η από το στένη κυρία Λέζινγκ και για το εργαστήριο αυτό έχουμε προσκαλέσει δύο προγνώμονες από το Ερευνητικό Κέντρο για την Ειρήνη Στοκχόλμης η κυρία Σίμπιλ Μπάουερ που είναι υπεύθυνη για θέματα εξοπλισμού και αφοπλισμού και η κυρία Μαλέτα βοηθός ερευνήτρια για το πρόγραμμα ελέγχου των πολίσεων όπλων. Επειδή το θέμα είναι ευρύ και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο αμέσως, κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Thank you very much to the chair and Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής που με προσκαλέσατε για να σας ενημερώσω για τον κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι εξαγωγέ όπλων. Είναι μια πρωτοβουλία που το Κοινοβούλιο παρακολουθεί εδώ και 20 χρόνια και που έχετε διδραματίσει ενεργό ρόλο και στον σχεδιασμό του ε, εργαλείου αυτού και στην εφαρμογή του και τον έλεγχο του πώ λειτουργήσε. Είναι χαρά μα λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ μαζί σα για να σα δώσουμε κάποια στοιχεία για το πώ λειτουργεί όλο αυτό. Θα κάνουμε την παρουσίαση στα δύο τμήματα και πριν ξεκινήσω ε, θέλω να πω δύο λόγια για το ε, ε, ίδρυμά μα, το Ινστιτούτο. Είναι σημαντικό όμω να θυμάστε και τη σχέση που έχουμε με το Κοινοβούλιο. Το Ίδρυμα εδρύθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο το 1966 για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ειρήνη και την ουδετερότητα στη Σουηδία. Ε, παραλάβαμε εντολή να παράσχουμε στοιχεία και να διερευνήσουμε τις συνθήκες για μια ειρήνη διαρκείας. Είναι λοιπόν ευρεία η εντολή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Εργαζόμαστε επί του θέματο εδώ και 50 χρόνια. Και επίση διευρύναμε το πεδίο εργασιών μα ε, στον τομέα των εξοπλισμών και του αφοπλισμού, καθώ και των συγκρούσεων και τη ειρήνη, για να δούμε ποια είναι τα αίτια των συγκρούσεων και τι μπορεί να απαιτεί σταθεροποίηση και η ειρήνη ή οι κλιματικέ αλλαγέ και οι προκλήσει στην ασφάλεια ε, από μια ευρύτερη προοπτική. Η Τζοβάνα θα ξεκινήσει δίνοντας σας μια γενική εικόνα κάποιους από τους αριθμούς που έχουμε συγκεντρώσει στο ΣΥΠΡΙ για την παραγωγή όπλων και τις μεταφορές τους και πώς αφορά αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα, τις πολιτικές και πρακτικές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ θα σας παρουσιάσω κάποιες δυνατότητες για να βελτιωθεί η κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον αποφασιστεί αυτό στο μέλλον. Τζοβάνα. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Τζοβάνα Μαλέτα, είμαι βοηθό ερευνήτρια στο ΣΥΠΡΙ και όπω ανέφερε η συνάδελφο, θέλω να σα δώσω πρώτα κάποιε λεπτομέρειε για το πώ τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία έχουν καθορίσει τον ε, ε, προπολογισμό του για τι αγορέ, μεταφορέ και πωλήσει όπλων. Και Ήθελα να σα δώσω κάποια στοιχεία για το πώ οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ τα τελευταία χρόνια στον τομέα του ελέγχου των ε, εξαγωγών όπλων έχουν παρουσιάσει διαφορέ τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντα από τι δαπάνε, τι αμυντικέ δαπάνε, βλέπετε από το διάγραμμα ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αμυντικέ του δαπάνε, την περίοδο από το 2008 στο 2016 ε, έχουν ε, περιορίσει τις δαπάνες τους. Τα δεδομένα που δίνει η βάση δεδομένων για τον αμυντικό εξοπλισμό δείχνει ότι υπήρξε μείωση από 240 ε, δις σε 229 το 2017. Την ίδια περίοδο ε, παρατηρούμε ότι τα κράτη-μέλη ε, στο σύνολό τους ε, των πωλήσεων από το 17% κατέβηκαν στο 15%. Ταυτόχρονα, κοιτάζοντας την κατάσταση, βλέπουμε ότι η τάση αυτή κάπως μεταβάλλεται και την περίοδο 2013-2017 οι αμυντικές δαπάνες άρχισαν και πάλι να μειώνονται. Συγκεκριμένα κατά 7% για όλα τα κράτη-μέλη μαζί. Και έχουμε και μια ομάδα κρατών, αυτούς που δαπανούν τα περισσότερα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, που το 2017 ήταν μεταξύ των 15 χωρών που ξόδεψαν τα περισσότερα παγκοσμίως βάσει των στοιχείων του ΣΥΠΡΙ. Και συνολικά φτάσαν το 10% του συνόλου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διαφορά μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών μελών, αυτών που δαπάνουν τα περισσότερα, βρίσκονται δηλαδή στο top 15 μαζί με, την, με τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία με 40 δις ευρώ το 2017 για να καταλάβουμε το πλαίσιο εντό το οποίο πρέπει να γίνει αναθεώρηση τη κοινή θέση. Πρέπει επίση να σκεφτούμε πώ η αμυντική βιομηχανία έχει ε, οργανωθεί τα τελευταία χρόνια βάσει των δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αμυντική βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 ε, είχε κύκλο εργασιών 97,3 δι. Και ξέρουμε βάσει των ίδιων ε, δεδομένων ότι η βιομηχανία αυτή έδωσε εργασία σε 500.000 εργαζομένους για την σύνθεση της βιομηχανίας αυτής να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ομάδα ε, εταιριών που δεσπόζουν στην αγορά και ακολουθεί και μια μεγάλη ομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίε είναι διάσπαρτε στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαιτέρω στα μεγαλύτερα κράτη όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία. Όπω όμω προανέφερα υπάρχουν κάποιε εταιρείε που είναι οι κορυφαίε. και βρίσκονται μεταξύ των 100 μεγαλύτερων εταιριών αμυντικού και στρατιωτικού εξοπλισμού βάσει των στοιχείων του ΣΥΠΡΙ. Ε, στο σχετική βάση δεδομένων του ΣΥΠΡΙ. Η βάση δεδομένων, ε, ε, η ιεραρχία της εταιρείας αυτής, της εταιρείας αυτής των πωλήσεών τους. Και αυτό που είδαμε είναι ότι μεταξύ του 2008 και 2016 ένας μέσος όρος 25 εταιριών που εδράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μεταξύ των 100 μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίω. Ταυτόχρονα όμως παρατηρήσαμε ότι στην υποεξέταση περίοδο το μερίδιο ως προς τις πωλήσει αμυντικού εξοπλισμού των ευρωπαϊκών εταιριών μέσα σε αυτές τις 100 πρώτες μειώθηκε και μειώθηκε από 31% περίπου στο, το 2008 σε 24% το 2016. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να είναι σοβαροί παράγοντες στον τομέα των εξαγωγών όπλων. Όπως βλέπουμε και από αυτή τη γραφική παράσταση, που βασίστηκε στα δεδομένα από την βάση δεδομένων για τις μεταφορές όπλων βλέπουμε ότι την περίοδο 2008-2017 το 2008 ήταν η χρονιά όπου άρχισε να ισχύει η κοινή θέση τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί έφταναν το 28% του συνολικού όγκου μεταφορών όπλων. Και εδώ έχουμε κάποιες χώρες που βρίσκονται στις υποτεστέσεις, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ε, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Από κοινού συνεισέφεραν σε αυτή την τάση και από το 2008 έφτασαν στο 23% του, συνόλου, του παγκόσμιου συνόλου. Για τη γενική αυτή εικόνα, καλό να αναφέρουμε και τι πρωτοβουλίε που αναλύθηκαν τα τελευταία χρόνια για να ενισχυθεί η συνεργασία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι πρωτοβουλίε που αναλύθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διακυβερνητικό επίπεδο. Και όπω θα ξέρετε, το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την άμυνα που αποτέλεσε τη βάση για την ε, ίδρυση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου πάλι το 2017 και όλοι ξέρουμε ότι η παραγωγή όπλων και το εμπόριο όπλων είναι εκτός της συνθήκης όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να λάβει κάποιο ρόλο σε αυτό το τομέα αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές της για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και με τον βιομηχανικό ανταγωνισμό. Πρότεινε λοιπόν μια δέσμη μέτρων με συνολικό στόχο να ε, ε, ενταθεί η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και να ενισχυθεί η, βάση των αμυντικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το Αμυντικό Ταμείο για πρώτη φορά ο προπολογισμό της Ένωσης θα συμβάλλει ώστε να χρηματοδοτήσει ε, δράσεις συνεργασίας στον τομέα των στρατιωτικών και για να ενισχύσει τις κοινέ στρατιωτικές δυνατότητες. Στο διακυβερνητικό επίπεδο πρέπει να σημειώσουμε το Δεκέμβριο του 2017 ξεκίνησε μια νέα μορφή συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία, που επέτρεψε σε πολλά κράτη-μέλη, όπω το επιθυμούν, να συνεργαστούν στο τομέα τη άμυνα και των στατιωτικών. Βεβαίω, η στρατηγική αυτονομία είναι απότερο στόχο όλων αυτών των προσπαθειών. Η ενίσχυση τη ενιαία αγορά ε, για τον αμυντικό εξοπλισμό, καλύτερε στρατιωτικέ δαπάνε, πιο εξορθολογισμένε όλα τα κράτη-μέλη και αντιμετώπιση των απειλών ασφάλεια στην ε, ε, γειτονία, στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, παραμένουν προκλήσει και για το μέλλον. Η πρώτη αφορά τι δυνατότητε των νέων κρατομελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιου τομεί, όπω την απόφαση για κάποια ε, προγράμματα ΠΕΣΚΟ, τις προτεραιότητες ε, των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ε, εάν θα παραμένουν τα κάποια εάν κάποια κρατημέλη θα παραμένουν υπεύθυνα για την έκδοση αδειών εξαγωγών όπλων. Όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη είναι τελικά υπεύθυνα για την υλοποίηση της κοινή θέση μέσω των εθνικών του συστημάτων. Τώρα, μετά από 10 χρόνια της ε, ε, ισχύω αυτής της θέσης, έχουν κληθεί να την αναθεωρήσουν για να δουν κατά πόσο είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των κριτηρίων της. Όπως θα ξέρετε, η κοινή θέση είναι ακρογωνίως λήθος όλων αυτών των προσπαθειών. Αλλά υπάρχουν και άλλα εργαλεία για το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναφέρω σύντομα, όπω η οδηγία για τι διακοινωτικέ μεταφορέ ή το εμπάργκο για τα όπλα και ένα φάσμα μέσων για τον έλεγχο ε, ε, στο εμπόριο των ε, διτής χρήσης προϊόντων. Δεν ήταν απλό να εγκριθεί η κοινή θέση. Το πρώτο βήμα προς την εναρπώνηση των πολιτικών ελέγχου για τις εξαγωγές ξεκίνησε το 1991. με την έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς για την ε, εξαγωγές όπλων το 2008 και φτάσαμε στην κοινή θέση. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι στα 10 αυτά χρόνια υπήρξαν κάποιες ε, περιπτώσεις όπου τα, οι πολιτικές των κρατών μελών στο τομέα των εξαγωγών όπλων ε, παρουσίασαν αποκλήσει, ιδίω σε περιπτώσει κρίση. Για παράδειγμα, κατά την Αραβική Άνοιξη, στο πλαίσιο το, ε, της σύγκρουσης στη Συρία ή της άρσης του εμπάργου στη Λιβύη. Και πιο πρόσφατα με τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Πράγματι, υπάρχει η κατηγορία η Κασία ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο παραβιάστηκε από τις ε, σαουδαραβικές δυνάμεις και αυτό υπονόμευσε την κοινή θέση. Το θέμα είναι κατά πόσον υπήρξαν εξαγωγές όπλων οι εξαγωγέ όπλων των ευρωπαϊκών κρατών προ τη Σαουδική Αραβία και των Αραβικών ε, Εμμυράτων ήταν ένα θέμα εδώ για το συνασπισμό. Ο συνασπισμός λοιπόν αυτός ε, φαίνεται ότι από το 2013 έως 2017 ε, ε, πήραν 50% παραπάνω όπλα από ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκά κράτη. Είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές τέτοιων όπλων προς τις χώρες αυτές η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ταυτόχρονα ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων που καλύπτω το 2016 δείχνει ότι υπήρξαν ε, αρνήσεις πωλήσεων προς τις χώρες αυτές βάσει του κριτηρίου 2 που υποτέθηκε ότι μπορεί να ε, παραβιάζεται και λήψη αυτού του 7 και υπήρξε ευρία συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί η κοινή θέση σε σχέση με αυτές τις εξαγωγές όπλων. Σε κάποιε περιπτώσει, οι συζητήσει αυτέ και η πίεση τη κοινή γνώμη οδήγησαν τα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε να ανακαλέσουν είτε να ακυρώσουν πωλήσει προ αυτέ τι χώρε, όπω οι κατοχώρε, η Βαλονία στο Βέλγιο και η Γερμανία. Κατά τα άλλα, άλλες χώρες αντιστάθηκαν στην πίεση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και η Γαλλία, και αυτό πυροδότησε μια σειρά από πρωτοβουλίες των πολιτών που κατηγόρησαν την κυβέρνησή τους για τις εξαγωγές αυτές. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να σταθεί η αναθεώρηση της κοινή θέσης. Οι αποκλήσεις της εξαγωγές όπλων υπήρξε ζήτημα μέσα σε αυτή τη δεκαετία και οι αποκλήσεις αυτές ε, θέτουν αμφιβόλο και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, ενισχύσει την ε, κοινή συνεργασία. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει και διαμεσολάβηση για να επιληθούν αυτές οι διαφορές. Εκεί θα μπορούσε να επικεντρωθεί αυτή η αναθεώρηση και τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο που θα σας παρουσιάσει κάποιες δυνατότητες Λοιπόν, τι κατάληξη θα μπορούσε να έχει αυτή η διαδικασία αναθεώρησης. Τονίζουμε ότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να είναι φιλόδοξη αυτή η αναθεώρηση. Η τελευταία αναθεώρηση που ξεκίνησε το 2011 και κατέληξε το 2015 είχε πολύ περιορισμένα αυτά αποτελέσματα. Και επειδή συμμετέχουν πολλοί που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και εμπλέκονται ενεργά σε αυτή την πολιτική, το κοινοβούλιο, η κοινωνία των πολιτών, οι διάφορες κυβερνήσεις και διάφορες άλλοι φορείς. Πρέπει λοιπόν αυτή η αναθεώρηση να γίνει χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να εκφραστούν. Πρώτη εναλλακτική είναι να γίνει μια διαδικασία εκτίμησης από ομοτήμους. Αυτό έχει γίνει για τα... την τεχνολογία διπλής χρήσης και έχει οδηγήσει αποτελέσματα. Αν υπάρχουν το μίσο που υπάρχει απόκληση απόψεων, καλό είναι να υπάρχει ε, ένα φόρουμ για να εκφραστούν οι λόγοι για αυτή την απόκληση και για να μπορέσει να γίνει εφικτή η εναρμόνιση. Πώς εφαρμόζεται η κοινή θέση της Ένωσης από τα διάφορα κράτη-μέλη. Αν το κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα, τι άδειε εξαγωγή όπλων δίνονται, αλλά και πολλέ διαφορέ επί τη διαδικασία. Πώ δηλαδή εφαρμόζονται τα κριτήρια μέσω εθνικών νόμων, μέσω πλαισίων αναφορά ή σε άλλε περιπτώσει δεν υπάρχει κανένα, καμία νομική βάση. Πώ λειτουργούν τα συστήματα σε κάθε κράτο μέλο, πολλές αποκλήσεις από κράτος σε κράτος. Ποια υπουργεία συμμετέχουν. Συμμετέχουν ε, με εξουσία συναπόφασης, ε, με δικαίωμα βέτο, ε, απλώς γίνεται διαβούλευση και αυτό έχει επιπτώσεις. Και τι μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Το ΣΥΠΡΙ έκανε μια μελέτη πραγματικά χρόνια τότε για την νορβηγική κυβέρνηση. Εξετάσαμε για παράδειγμα το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο, τις μεθόδους και τις πηγές που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για αυτήν την αξιολόγηση. Και υπήρξαν πολύ έντονες διαφορές. Θα στείλει στην πρεσβεία σου ένα τρισέλιδο ερωτηματολόγιο ή μία μόνο ερώτηση. Και από τι πηγές θα πάρεις πληροφορίες. Για να απαντήσεις ε, τα διάφορα ερωτήματα που έχεις θέσει. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα τη γενικότερη πολιτική Άμα δει τι λεπτομέρειες τη εφαρμογής της πολιτικής, μπορείς να εξαγάγει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που οδηγούν στην αναρμόνιση. Και έτσι μπορεί να γίνει και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Μέσω αυτή τη διαδικασία αποτίμηση ομοτήμων δημιουργήσει ένα φυσιολογικό φόρουμ για ανταλλαγέ απόψεων. Υπάρχουν τακτικέ συνεδριάσεις, αλλά δεν υπάρχουν πολύ άτυποι τρόποι με τους οποίους οι αρμόδιοι για τη χορήγηση τέτοιων αδειών μπορούν να ανταλλάξουν απόψει Και πολύ λιγότερο και αυτοί οι οποίοι ε, συμμετέχουν μετά στην παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινή θέση. Πολλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει, να γίνουν μάλλον. Κάτι άλλο που είναι το επόμενο πώς υποβάλλονται και εκθέσεις για το τι γίνεται. Και εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα συστήματα. Όταν προτίμαζα αυτή την παρουσίαση, εξέτασα μία μελέτη που είχα κάνει με έναν συνάδελφο στο ΣΥΠΡΙ το 2004. Συγκρίναμε τις διάφορες μεθόδους ε, συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τις εθνικές εκθέσεις και για τις ε, συμβολές στην ετήσια έκθεση της Ένωσης. Διάφορα θέματα που υπήρχαν τότε εξακολουθούν να εκκρεμούν και τώρα, 14 χρόνια κατόπιν. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στο σχεδιασμό των θεμάτων αυτών. Δεν υποβάλλουν πλήρε εκθέσει για την ετήσια έκθεση όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση επίση. Μπορεί να βελτιωθεί και η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των στοιχείων. Για παράδειγμα, πληροφορίε για το ποιοι είναι οι τελικοί χρήστε, για ποσότητε εξαγωμένων όπλων. Μερικά από τα μεγάλα κράτη-μέλη δεν δίνουν όλα του τα στοιχεία για τι εξαγωγέ όπλων. Το είχαμε θίξει πριν από 14 χρόνια. Υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε, να δούμε και τι πληροφορία, πληροφόρηση και στοιχεία έχουν ε, οι επιχειρήσεις που εξάγουν τα όπλα, οι πελάτες. Ε, ε θα μπορούσε να ήταν, ε, για παράδειγμα, μια απλή ενέργεια να του στείλουμε πίσω την έκθεση, αν είναι λυπής. Και κάτι άλλο. Η σημερινή μας έκθεση δημοσιεύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 18 αλλά καλύπτει την κατάσταση του 16. Μάλιστα ήταν η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, κάτι άλλο. Πώς θα βελτιωθούν αυτές οι εθνικές εκθέσεις. Στην κοινή θέση αναφέρεται ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκδίδουν και αιτήσιες εκθέσεις. Και είναι πολύ διαφορετικές αυτές από χώρα σε χώρα. Πόσο συνολικές είναι, πόσο έγκαιρα βγαίνουν, τι ποσότητα και ποιότητα περιέχουν. Δεν θα πω περισσότερα. Αλλά κατόπιν αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ. Επίσης, και η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ κρατών μελών μπορεί να βελτιωθεί. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Μετά την τελευταία διαδικασία επανεξέτασης υπάρχει μια βάση δεδομένων όπου μπορεί να γίνει ανταλλαγή στοιχείων αλλά θα μπορούσαν να στέλνουν περισσότερα στοιχεία. Για παράδειγμα, παρελθούσες περιπτώσεις όπου έχουν εκτραπεί τα όπλα και επίσης αν ένα κράτος μέλος αναστέλει ή ακυρώνει μία άδεια εξαγωγής. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών. Και αυτό θα βοηθούσε και τις αρχές που παρακολουθούν μετά την εφαρμογή του νόμου. Τα οχτώ κριτήρια και όλες, ε, όλα τα άλλα κείμενα είναι παλιά, 10 και 20 ετών. Θα πρέπει να εξετάσουμε ευρύτερα αυτά τα οχτώ κριτήρια και να δούμε, είναι ακόμη κατάλληλα, μπορούν να τροποποιηθούν. Και το ίδιο και για τον οδηγό χρήσης χρήσιμο, αλλά θα μπορούσε και αυτός να ενημερωθεί, να γίνει πιο ευανάγνωστος, να αναφέρει τι πηγές του περισσότερο. Να μην ε, επιδιώξουμε λοιπόν ελάχιστες μόνο βελτιώσει, Να θέσουμε το ερώτημα, εάν τα φτιάχναμε από την αρχή, έτσι θα τα φτιάχναμε. Σημαντική ερώτηση. Και ένα από το θέμα για τα κριτήρια. Ήδη αναφέρθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο η διαφορά μεταξύ μιας ε, προσέγγισης που βασίζεται σε αρχές, όπου εξετάζει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα, ή αν εξετάζεις μόνο από λειτουργική άποψη, εάν ένα συγκεκριμένο όπλο δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να τα ξαναδούμε αυτά. Και επίση ε, η εκτροπή προ άλλου χρήστε, Διότι εάν διαπιστώσουμε ότι πάνε κάπου αλλού τα όπλα μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να ακυρώσουμε την άδεια εξαγωγής ή ε, σε άλλες περιπτώσεις απλώ λαμβάνεται υπόψη. Θα μπορούσε αυτή η εκτροπή σε άλλο τελικό χρήστη, θα μπορούσε να οδηγεί σε ακύρωση της εξαγωγής όπλων. Τώρα για τα όπλα διπλής χρήσης. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των διαδικασιών εφαρμογής και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις αν υπάρξουν ε, παραβιάσεις. Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και για τις ε, εξαγωγές όπλων, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα εθνική. Αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι διαφορές, γιατί έχει τεράστιες επιπτώσεις και για τις εταιρείε και για τα άτομα. Και επίση, τι πόρους διαθέτουν οι αρχέ αστυνομία. Θα μπορούσαμε να αποφεληθούμε από την πύρα για τα προϊόντα διπλής χρήση. Να δούμε δηλαδή πόσε άδειε, συγγνώμη, πόσοι δουλεύουν σε κάθε υπηρεσία χορήγηση αδειών και εφαρμογή των αποφάσεων. Γιατί οι παλιότερε μελέτες είχαν, ε, κατέληξαν σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα όταν ε, μας ε, όταν τους ρωτήσαμε ποια είναι η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν για να κάνουν τη δουλειά τους, ε, οι περισσότεροι μας είπαν ότι δεν έχουμε επαρκείς πόρους και επαρκές προσωπικό. Επίσης, πρέπει να συμμετέχουν περισσότερα τα ενωσιακά όργανα στη, για την παροχή και εξέταση των πληροφοριών. Ιδιαίτερα τα μικρότερα κράτη-μέλη πολλέ φορέ ε, έχουν μεγάλε δυσκολίε. Δεν έχουν αρκετά ευρύ δίκτυο πρεσβειών, για παράδειγμα, στο εξωτερικό για να λάβουν πληροφόρηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και αντιπροσωπείε τη Ένωση για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Η Τζοβάνα το ανέφερε ήδη. Το καθεστώς ε, ελέγχου των εξαγωγών όπλων είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένο. Όχι μόνο τα τρία θεσμικά όργανα, αλλά και διάφορε υπηρεσίε ε, εντό αυτών των οργάνων. Θα έπρεπε να συνδυάσουν περισσότερο την εργασία του. Γιατί στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει παρόμοιο επίπεδο κατακαιρματισμού. Πολλά θέματα τα αντιμετωπίζουν ε, ε, μόνο σε μία υπηρεσία σε ένα κράτος μέλος, ενώ στην Ένωση είναι πολύ διαφορετικές και πολλές οι υπηρεσίες που ασχολούνται. Ορίστε, σας δώσαμε και διάφορα στοιχεία και σας έχουμε και διάφορα κείμενα εδώ και δημοσιεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Μαλέτα και την κυρία Μπάουερ για, αυτή την πολύ, για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και όλα τα σχολεία τους σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ε, εφαρμογής της κοινή θέση. Στρέφομαι στην κυρία Λέζινγκ που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη πέρυσι είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και πολλά από τα ουσιώδη προβλήματα έκτοτε δεν έχουν επιληθεί. Δεν έχει προχωρήσει καν η λύση τους. Λοιπόν, να ασχοληθώ με το εξή. Είπατε σε διάφορα σημεία η κοινή θέση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά. Ακούγεται πολύ και στο Κοινοβούλιο αυτό. Όταν ακούω τέτοια πράγματα στην Επιτροπή ή στο Κοινοβούλιο ανησυχώ. Γιατί πολλές φορές έχω την εντύπωση και το φόβο ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση της εφαρμογής της κοινή θέση, αλλά πολλές φορές στόχος είναι η αποδυνάμωση της. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να επανεξεταστούν τα διάφορα κριτήρια Ανησυχώ ιδιαίτερω. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο και πάλι, να ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση του περιεχομένου τη κοινή θέση και όχι απλώ να συζητήσουμε την εφαρμογή τη, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω τη δική σας παρουσίαση ως προσπάθεια για μια καλύτερη και πιο αυστηρή εφαρμογή της κοινής Και γι' αυτό το λόγο ορισμένα κριτήρια θέλετε να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Οπότε το ερώτημα μου είναι πώς θα αποφύγουμε αυτή η πανεξέταση να πάει προς την άλλη κατεύθυνση. Εάν συζητήσουμε το περιεχόμενο της κοινή θέση, τότε ίσως κάποια κριτήρια, για παράδειγμα η συμβατότητα με την αναπτυξιακή πολιτική, μήπως θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν αυτά τα κριτήρια αν τα επανεξετάσουμε. Αναφερθήκατε στα όπλα ή στα προϊόντα διπλής χρήσης. Νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο σημαντικός αυτός ο τομέας. Οπότε, μήπως μπορείτε να μα μιλήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα, να μας πείτε μάλλον πιο συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις και με τι τρόπο θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο, δεν ε, έχει να κάνει μόνο με εξαγωγές. Για παράδειγμα, τι διαρθρωτικές βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε εντός της Ένωσης, ούτως ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία αυτό ο τομέα των προϊόντων διπλής κρίσης και κατόπιν οι πόροι και το προσωπικό. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Την πολιτική του βούληση να εφαρμοστεί αποτελεσματικά αυτή η κοινή θέση. Γιατί η επάρκεια πόρων για να γίνει αυτό είναι φυσικά καθήκον των κρατών μελών. υπάρχουν τουλάχιστον ε, ελάχιστες απαιτήσει που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε ούτω ώστε κάθε έκθεση κράτους μέλους να περιέχει τουλάχιστον ορισμένα για να μην έχουμε να διαβάσουμε 20 ε, τόσο διαφορετικές εκθέσεις που είναι δύσκολο να τις συγκρίνεις μετά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να εναρμονίσεις αυτές τις εκθέσεις αλλά κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές δεν θα βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένες, ελάχιστες απαιτήσει. Μία, δύο, τρεις. Τώρα λέτε ότι πρέπει να βελτιωθεί η νομική πλευρά της κοινή θέση για να γίνει ευκολότερη η εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να μας γίνει τι θέλετε. Κατόπιν. Κάτι που δεν έχουμε αναφέρει ακόμη. Υπάρχουν ε, μεγάλες προκλήσεις όπως έχουν τώρα οι προϋποθέσεις που θέτουμε. Μετά υπάρχουν και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα της Ένωσης. Το EDIDP Σκεφτήκατε με τι νέες συνθήκες πρέπει να γίνει. Σε σχέση και με τη νέα διευκόλυνση ειρήνης. Ποιες πρέπει να είναι οι προποθέσει που πρέπει να θέσουμε για τους τελικούς χρήστες. Μήπως αυτά θα πρέπει να το βγάλουμε το edit και από τη διευκόλυνση Ειρηνή και να τα έχουμε σε ένα ενοποιημένο σύστημα ελέγχου. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις μου. Thank you. I... Ευχαριστώ πολύ ο λόγος. Βαλέρο. Ε, χαίρομαι που έχουμε εδώ πέρα εκπροσώπους του ΣΥΠΡΙ. Ε, πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι για το ΣΥΠΡΙ, το οποίο το στηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Το ξεκινήσαμε πριν από δεκαετίες και βλέπω ότι πια έχει καταφέρει να εδρεωθεί στη συνείδηση όλων. Αν μπορούσατε να μας στείλετε και τι διαφάνειε σας γραπτό θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο. Η Σαμπίνε ε, ή είπε ότι θα ήταν χρήσιμο να διευρύνουμε τη συζήτηση έτσι ώστε να εδρεωθεί και η ίδια εκείνη θέση. Όπως είπε η Σαμπίν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση ε, να μειωθούν οι απαιτήσει. Έχουμε μια κοινή θέση η οποία είναι αξιόλογη. Και επίσης έχουμε και το δεύτερο κριτήριο των βασικών αρχών και της, ε, της λειτουργικής εστίασης. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει αυτή η προσέγγιση. Γιατί η τάση είναι η εναρμόνιση να περιοριστεί ε, και να γίνει λιγότερο αυστηρή. Γίνεται προσπάθεια κωδικοποίηση των πρακτικών ε, μέσω συμμετοχής πολλών ε, εμπλεκομένων και ο, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα τελικά είναι ότι ο νόμος αντικατοπτρίζει, προσπαθεί να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα αντί να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή ο νόμος ε, να είναι αποτέλεσμα μιας ε, συζήτησης και της συγκεκριμένων κριτηρίων. Θέλουμε δηλαδή στο μέλλον να ε, βελτιώσουμε τα κριτήριά μας, όχι να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα που εξελίσσεται. Ποια είναι η δική σας γνώμη, ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι για το μέλλον, πόσο σοβαροί είναι αυτοί οι κίνδυνοι στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την τελική χρήση των πόρων, θα πρέπει να προγραμματίσουμε αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στους ελέγχους μας. Τι νόημα έχει μια κοινή θέση στα χαρτιά όταν στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται μέσω ελέγχου και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει σε όλο τον κόσμο. Χωρίς ελέγχους, χωρίς επιθεωρήσεις δεν θα προχωρήσουμε. Τα κράτη-μέλη τα οποία συνεχίζουν να πολλούν στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα θα πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν σε ζώνες ε, εμπόλεμες όπως η Εμένη. Αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι δεν αρκούν. Πώς θα καταφέρουμε τα κράτη-μέλη να σεβαστούν αυτές τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ. Κύριο Σκύλα, έχετε το λόγο. Πολύ χρήσιμες και πρακτικές συμβολές σας. Είπατε ότι συχνά σε περιπτώσεις σημαντικών κρίσεων όπως την Ιεμένη, τη Συρία, η κοινή θέση συχνά αγνοείται, υπά και παραβιάζεται. Έχετε να μας ε, πείτε κάτι για το πώς θα μπορούσαμε να προετοιμαστούμε για κάποιες μελλοντικές κρίσεις τέτοιου τύπου. Και μετά το θέμα, το παντοτινό θέμα της ανεπαρκούς εναρμόνισης και μάλιστα και σε εθνικό επίπεδο πολλές φορές υπάρχουν διαφορές ε, μέσα στην ίδια χώρα αλλά και επίσης σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση της κοινή ε, Εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε αλλά δεν βλέπω μια καλή λύση. Οπότε τελικά το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Μόνο αν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προβαίνουν σε πιο αυστηρούς ελέγχους, πιο αποτελεσματικούς ελέγχους των εθνικών συστημάτων θα τα καταφέρουμε. Είπατε ότι η έλεγχοι εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατακαιρματισμένοι και βέβαια εδώ παίζει ρόλο και η χρηματοδότηση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει να εναρμονίσει και να εφαρμόσει ευρωπαϊκούς ελέγχους, σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα και το Κοινοβούλιο έχει να παίξει το ρόλο του και σε αυτό. Επίσης, γίνεται μια, μια προειδοποίηση για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε εμπόριο όπλων και εξαγωγές. Υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, πιο αποτελεσματικά μέτρα για να έχουμε τέτοιου είδους προειδοποίησεις, να λαμβάνουμε τέτοιου είδους προειδοποίησεις έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τις πρώτες ερωτήσεις, ο λόγος ξανά σε εσά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Οι ερωτήσει πράγματι ήταν ενδιαφέρουσε. Θα απαντήσω σε μερικέ και θα δώσω το λόγο και στη συνάδελφό μου για να απαντήσει στις υπόλοιπε. Αν υπάρχει κίνδυνο με την, με την συζήτηση των κριτηρίων σε μια πιο ευρεία συζήτηση, σε, μια πιο, σε ένα πιο ευρύ κύκλο. Πάντοτε υπήρχε αυτό ο κίνδυνο και εξακολουθεί να υπάρχει, όπω υπάρχει και ο κίνδυνο στην εφαρμογή των κριτηρίων. Γιατί κάποια από αυτά τα κριτήρια ε, ορίζονται με έναν τρόπο τόσο ευρύ που μπορούν να παρεμεινευθούν και να εφαρμοστούν με διαφορετικούς τρόπους. Αν επιλέξουμε να αποσαφηνίσουμε την διατύπωση, τότε ο κίνδυνος αυτός θα μειωθεί και πλέον τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα ενδεχομένως να αναφέρουν ποια είναι η δική τους ερμηνεία για κάθε κριτήριο. Αυτή η διαδικασία θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμη. Αυτή η αρχική διάκριση ανάμεσα στο τι πρέπει να λάβετε υπόψη και ενδεχομένω να το απορρίψετε και τι θα πρέπει να εφαρμόσετε ρητά ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνει και χρήσιμο. Ε, το ε, Κριτήριο της ε, εκτροπής επίσης είναι, συγγνώμη, της ανάπτυξης, το αναπτυξιακό κριτήριο ληφθεί υπόψη, θα είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν του έχει δοθεί τόση έμφαση στο παρελθόν. Αυτοί οι οποίοι εξετάζουν θέματα αναπτυξιακά πρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση γιατί αλλιώς το κριτήριο αυτό παραμερίζεται. Ενδεχομένως είναι ανιαρό να εξετάζει κανείς τις διαδικασίες, αλλά όταν το κάνει τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ στην πράξη, διότι περνάμε από την θεωρία στην πράξη με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τις διαδικασίες θα πρέπει να τις δούμε ε, και να τις εξετάσουμε στενά και προσεκτικά. Επίσης, έχουμε και τη συνθήκη εμπορίας όπλων, την οποία δεν είχαμε δεν διαθέταμε όταν υιοθετήσαμε τα οκτώ κριτήρια για τον κώδικα δεοντολογίας. Οπότε έχουμε πλέον μια ελάχιστη παγκόσμια προδιαγραφή, την οποία είναι αδύνατον πλέον να αγνοούμε. Ρωτήσατε επίσης τι μπορεί να γίνει για να βελτιώσουμε την εφαρμογή της κοινή θέση και να αποφύγουμε ε, τη χαλαρότητα σε περιπτώσεις κρίσεων. Ε, η συνθήκη εμπορίας όπλων είναι σημαντική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τη λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της μαζί με τα κριτήρια. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι διεθνείς παίκτες. Δεν μπορούμε να προωθούμε κριτήρια σε άλλους και να θέλουμε να τα εφαρμόζουν και να, να, και να μην τα παίρνουμε στα σοβαρά εμείς. Οπότε αυτά που κηρύττουμε στους άλλους πρέπει και εμείς οι ίδιοι να τα πράττουμε. Μετά τέθηκε ένα θέμα σε ό,τι αφορά τους πόρους και τη χρηματοδότηση. Δεν αφορά μόνο τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορεί να βοηθήσει. Προφανώς η, τα ποσά κινητοποιούνται σε εθνικό επίπεδο κυρίως. Αλλά ε, είναι ηρωνικό και στις εξαγωγές όπλων και στον εξοπλισμό διπλής χρήσης υπάρχουν, ότι υπάρχουν ε, πολλά διεθνή προγράμματα αλλά όχι ένα πρόγραμμα για την άδειε, για παράδειγμα εμπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στην διαδικασία ανα, ε, αναθεώρησης ή αξιολόγησης μάλλον θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποιο κείμενο έτσι ώστε να αναγκαστούν τα κράτη-μέλη να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την υλοποίηση των κριτηρίων της κοινή θέση. και να συμπεριλάβουμε και μια ε, διαδικασία αξιολόγηση από ομοτήμου που θα περιλαμβάνει και το πόσο τι ποσά ε, δαπανώνται για την ε, εφαρμογή των κριτηρίων. Εκεί θα φαινόταν ότι ορισμένε χώρε υποχρηματοδοτούν. Ε, για τι εκθέσει δεν νομίζω ότι είναι επιθυμητό να εναρμονιστούν οι εθνικές εκθέσει. Γιατί νομίζω ότι έτσι θα χάναμε πολλές πληροφορίες. Πολύ δε περισσότερο που το κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να θέλει να εξετάσει συγκεκριμένα θέματα. Και υπάρχουν και εθνικά κριτήρια, εθνικέ διαδικασίε, εθνική νόμοι που πρέπει να, τύχουν σεβασμού. Όμω, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην κοινή θέση κάποια ελάχιστα κριτήρια και ελάχιστε προϋποθέσεις για τι εκθέσει. Αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ποσότητες, Συγγνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε θα πρέπει να περιλαμβάνουν ε, ορισμένα ελάχιστα βασικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τι ε, άδειε που ε, δόθηκαν, τα ποσά κλπ. Και επίση κάποιε ε, ε, ελάχιστες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τα εθνικά κοινοβούλια να αξιολογήσουν την κατάσταση γιατί μόνο τα αριθμητικά στοιχεία δεν αρκούν. Θα πρέπει να δούμε τι τύποι ε, όπλων πουλήθηκαν, ποιος ήταν ο τελικός ε, αγοραστής κλπ. Όλα αυτά ίσως είναι οι ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε εκθέσεις. Έλεγχη στους, για την τελική χρήση. Εδώ είναι ένα θέμα που τα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη, έχουν κάνει βήματα πρόοδου, αλλά αυτό δεν έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γερμανία, παράδειγμα, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα για τον έλεγχο τελική χρήση. Του πήρε κάποιο χρόνο γιατί χρειάστηκε να κάνουν και αλλαγές στο νομικό καθεστώς τους. Ε, όταν γίνεται μια σύμβαση με μια χώρα θα πρέπει να περιλαμβάνονται ε, νομικές διατάξεις, ε, για παράδειγμα που υποχρώνουν αυτή τη χώρα που αγοράζει να τα χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο τρόπο. Χρειάζεται όμω κάτι τέτοιο να διευρυνθεί, ένα τέτοιο σύστημα να εφαρμοστεί από άλλε χώρε και ενδεχομένω θα μπορούσε να ενταχθεί στην ε, κοινή θέση. Σε ό,τι αφορά την βελτίωση της εφαρμογής, ένας από τους ε, τρόπους για τη βελτίωση και για την βελτίωση συνεργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών. Ήδη γίνονται ανταλλαγές για την παράνομη χρήση, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις ε, πληροφορίες που μπορούν να ε, τοποθετηθούν σε μια κοινή βάση εξαιτία των κανόνων ε, προστασίας των δεδομένων κλπ. Αν είχαμε ένα φόρουμ που θα συνεδρίαζε μια φορά το μήνα στη Βρυξέλλες για παράδειγμα, θα μπορούσαν να γίνουν ανταλλαγές σε ό,τι αφορά αυτές τις δραστηριότητες και να βελτιωθεί η εφαρμογή των κανόνων για την χορηγήση αδειών εξαγωγής. Και εδώ βέβαια έχουμε ένα θέμα πόρων και χρηματοδότησης, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ένα τέτοιο φόρουμ. Τα Δίνω το λόγο τώρα στην Τζοβάνα να απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα. Uh, we, we close up... Πριν ολοκληρώσουμε, να σχολιάσω και εγώ τις παρατηρήσεις που έγιναν για τις πιθανές συνέπειες που θα έχει δημιουργία του Ταμείου για την άμυνα στις εξαγωγές όπλων. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά χωρίς απάντηση. Διότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται οι εξελίξεις οι ίδιες. Αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει είναι να γίνονται πολλές προσπάθειες, να συγκεντρωθούν πόροι για κοινά προγράμματα στον τομέα της τακτικής έρευνας και να συνδυαστούν οι δυνατότητες στην άμυνα. Όμως τα κράτη-μέλη παραμένουν καθήλυνα αρμόδια για την ε, χορήγηση αδειών στις εξαγωγές. Οπότε υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις στο πώς εφαρμόζεται εκείνη η θέση. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες για να συσταθεί μια επιτροπή και να αξιολογεί τις προτάσεις για σχέδια. Νομίζω δεν έχουν διοριστεί ακόμη οι επιρρογνώμονες, δεν έχει γίνει επιλογή Θα είναι όμως κάποιο είδους επιτροπή διοντολογίας για να μπορεί να ελέγξει το κατά πόσον τα προγράμματα αυτά σέβονται τη διοντολογία ή όχι. Έχει και κάποιες άλλες ε, δράσεις υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μετά το 2020. Πάντως, είναι λίγο νωρίς για να υπολογίσουμε Πώ θα επηρεαστεί η χορήγηση αδειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποιε σύντομε παρατηρήσει για την Ιεμένη λόγου χάρη. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν συγκεντρώνα στοιχεία για τη χορήγηση αδειών και κοίταζα κάποιε περιπτώσει από το παρελθόν, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ε, στην ιστορία των κρατών μελών κάτι τέτοιο. Μια κρίση προκύπτει και η συνεκτικότητα της κοινή θέση κλονίζεται. Αυτό το είδαμε και στην Ιεμένη και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Ίσως τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου όταν εξετάζουν τις άδειες που χορηγούν και υπάρχουν και πολλά διδάγματα από το παρελθόν. Το είδαμε στη Λιβύη, την Αραβική Άνοιξη, την Συρία. Ίσως από τις πρώτες στιγμές που υπήρξαν αφισβητούμενες πολύ όπλα προς την Μέση Ανατολή, ε, τη δεκαετία του 90 λοιπόν τα ξεκίνησαν οι πρώτες κοινέ προσπάθειες, να είναι ένας τρόπος να δούμε τι έγινε τότε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τις δυο σας για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τις τόσες λεπτομέρειες που μας δώσατε για αυτό το σημαντικό τομέα εργασίας του Κοινοβουλίου. Έχω δεχτεί το αίτημα, εάν μπορείτε, να μας δώσετε και αντίγραφα των διαφανειών. Έστω και ηλεκτρονικά μετά το πέρας της συνεδρίασης. Για να έχουμε μια επενθύμηση των πληροφοριών που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα το πρωί μαζί μας για αυτή την τόσο ε, ενδιαφέρουσα συνεισφορά στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Και τώρα θα παραδώσω την Προεδρία στην Πρόεδρο της Επιτροπής μας. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ. Colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Καλημέρα κύριε και κύριοι. Να συγχαρώ την αντιπρόεδρό μας Claire Moody για τον έγκαιρο χρόνο με τον οποίο την κατάλληλη στιγμή για ολοκλήρωση της ζήτησης και Uh-huh. Give them a bit of time to get settled. I'm sorry. Mm-hmm. Okay, we, we wait. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα για να... Ε, τακτοποιηθούμε. Okay, Λοιπόν, λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο θέμα στην ημέρηση διάταξη είναι το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για το EDIDP, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Άμυνα και τη Βιομηχανική ε, Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ο συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Μιρτσέα Πάσχου. Οπότε παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η Ήτρε ενέκρινε το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Ψήφισαν και σε δύο εβδομάδε στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε για την έκθεση. Έγινε πολύ έντονη συζήτηση στον τριμερή διάλογο. Τέσσερις γύροι, αν θυμάμαι καλά. Ο τελευταίο διήρκησε περισσότερο από τους προηγούμενους. Και τελικά λύσαμε όλα τα προβλήματα. Το Κοινοβούλιο επέμεινε ιδιαίτερα σε διάφορα σημεία που θα αναφέρω. Μετά υπήρξαν μόνο δύο αντιδράσεις στο αποτέλεσμα της συζήτησης από το Συμβούλιο. Η Κορεπέρα έκανε δύο προτάσεις. Η μία είναι δεκτή, η άλλη όχι. Τελικά το Συμβούλιο ενέκρινε το κείμενο και το ενέκρινε και η με ευρία πλειοψηφία σήμερα το πρωί. Λοιπόν, διάφορα σημεία ετέθησαν και ήταν στη θέση μας και τα συζητήσαμε με το Συμβούλιο, κυρίως με το Συμβούλιο. Το πρώτο θέμα ήταν οι επιλέξιμες ενέργειες. Ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν η φόρμουλα 3 συν 3 για, τα επιλέξιμα, για τους επιλέξιμους ομίλους εγκρίθηκε αυτό. Η συγχρηματοδότηση για τα, από τα κράτη-μέλη των στοιχείων του κόστους που δεν καλύπτει το πρόγραμμα και τα χρηματοδοτικά όργανα δεν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αλλά από ό,τι κατάλαβα θα υπάρξει μια νέα διατύπωση που θα αποδεχθεί αυτά τα χρηματοδοτικά όργανα. Κατόπιν κάποια υποχρέωση είχε αναλυφθεί από τις χώρες, τα κράτη-μέλη, να ενισχύσουν τις συνοδευτικές τεχνολογίες. Και έχουμε από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη μία δήλωση πρόθεσης. Αυτό είναι καινούργιο. συζητήθηκε επί μακρόν και αποδέχθηκαν τη δική μας διατύπωση. Ο εξοπλισμός και τα τεχνολογικά προϊόντα που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο δεν θα πρέπει να ενισχύονται από το πρόγραμμα. Δηλαδή, οι απογορευμένες ενέργειες με βάση το διεθνές δίκαιο είναι αυτές που περιέχονται στη γνωμοδότηση ΑΦΕΤ ΣΕΝΤΕ. Αγωνιστήκαμε πολύ για το σημείο αυτό, αλλά τελικά κερδίσαμε σε αυτό το σημείο. Κάτι άλλο που προέβαλε το Κοινοβούλιο είναι οι επιλέξιμες, ε, οι επιλέξιμοι φορείς. Εμείς θέλαμε να έχουμε πολύ αυστηρά κριτήρια για το θέμα αυτό και υπήρξε διαφορά απόψεων με, μεταξύ των ε, φορέων που ελέγχονται από τρίτες χώρες αλλά που ε, είναι εντός και εκτός της Ένωσης. Για, αυτές, για αυτούς τους φορείς που είναι εντός της Ένωσης θα ελέγχουμε το δομέα διοίκηση, δεν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες προφορίες και δεν θα υπάρχει ιδιοκτησία των αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς τους. Για τις επιχειρήσεις που είναι εκτός της Ένωσης μπορούν, είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και σε ενέργειες, αλλά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα και υφίστανται παρόμοιους περιορισμούς. εάν δεν είναι κρίσιμη η συμβολή τους στην ε, αλυσίδα παραγωγών, ε, συγγνώμη, ε, παραγωγής προϊόντων, δεν θα χρηματοδοτούνται από το Edit. Και τον τελικό έλεγχο θα το κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτή ήταν η θέση του Συμβουλίου και υποχρεωθήκαμε να το δεχθούμε. Εμείς ε, θέλαμε ακόμη πιο αυστηρούς ελέγχους, αλλά εφόσον ικανοποιεί αυτή η κατάσταση στα κράτη-μέλη, συμφωνούμε. Επίσης θέλουμε να συμπεριληφθούν σε αυτή την αλυσίδα παροχής, σε όλη την Ένωση, οι μικρομεσαίες και οι εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχαμε προβάλει ιδιαίτερα στην υποεπιτροπή μας. Τώρα η δομή για τα μπόνους. Η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη ε, διαρθρωμένη συνεργασία, θα πάρει ένα 10% επιπλέον. Οι μικρομεσαίες θα πρέπει να συμμετέχουν με 10% του συνολικού προπολογισμού. Επιπλέον μπόνους για τη συμμετοχή μικρομεσαίων θα δίδεται. Οι εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να λάβουν το 10% και το συνολικό μπόνους πρέπει να φτάνει μόνο μέχρι το 35% των ε, επιλέξιμων δαπανών. Γιατί αλλιώ θα υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών και τελικά δεν θα πηγαίναμε πουθενά. Ο προπολογισμό, βέβαια, ήταν ε, το σημείο που έγιναν οι περισσότερε διαπραγματεύσει. 500 εκατομμύρια για το 19 και το 20. 60% του οποίου θα έρθει από την αναδιανομή ε, των υπαρχόντων προγραμμάτων και 40% από το μη δαπανηθέν ε, περιθώριο του υπάρχοντος πολιτούς πλαισίου. Εκεί έγινε η μάχη μεταξύ 60 και 40. Γιατί ήταν 85 και 15. Αυτό το επιτύχαμε την τελευταία στιγμή. Και το Συμβούλιο τελικά υποχώρησε. 60% αναδιανομή από άλλα ενωσιακά προγράμματα και 40% από το παρόν ε, πολιτές πλαίσιο από το μη χρησιμοποιηθέν περιθώριο. Το Συμβούλιο βέβαια μας είπε, όπως και η Επιτροπή, ότι δεν ξέρουμε τι τελικά ποσά θα μας μείνουν. Τι μπορεί να μας προκύψει. Και θα είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη εντός του υπαρχόντος πλαισίου επιπλέον ε, πόρους. Αλλά τελικά καταφέραμε να τους πείσουμε ότι 40% θα πρέπει να προκύψει από αυτό το περιθώριο. Δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας και ιδιοκτησία γενικότερα. Αναφέρθηκε και αυτό. Υπάρχει ε, ε, μια δυνατότητα να επιτηρεί το πρόγραμμα οικομισιών Οποτεδήποτε υπάρξει μεταφορά διοκτησία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή, χωρί αυτό να περιορίζει τι δυνατότητε των κρατών μελών να εξάγουν όπλα. Επ' αυτό βεβαίω τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να καταλήψουν την ε, αρμοδιότητά τους. Εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει το πρόγραμμα με απευθείας ε, οικονομική διαχείριση. Αυτή ήταν η γνώμη μας. Άλλοι θέλανε την άλλη δυνατότητα που θα μας έδινε περισσότερο έλεγχο αλλά ε, για τα επόμενα δύο χρόνια έτσι θα επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αν αφήσουμε στα χέρια της Επιτροπής με τη διαδικασία απευθείας οικονομικής διαχείρισης. Με εφαρμοστικές πράξεις για το, την επόμενη διετία αναφέραμε τις κατηγορίες ε, αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογιών για να υπάρξει ευρύ πεδίο για τεχνολογική καινοτομία. Θα υπάρχει μια επιτροπή που θα βοηθάει την επιτροπή για την ε, εφαρμογή του προγράμματος και τον ε, Ευρωπαϊκό Φορέα Άμυνας και χαιρετίζω την παρουσία του Χόρχε που είναι επικεφαλής, ο κύριος Χόρχε Ντομέκ που είναι επικεφαλής του φορέα. Ο κύριος λοιπόν Χόρχε Ντομέκ θα παρακολουθεί ως παρατηρητής της εργασίας αυτής της Επιτροπής. Γιατί όπως ε, επιχειρηματολογήσαμε υπάρχει πολλή τεχνογνωσία και πείρα στον Ευρωπαϊκό Φορέα Άμυνας που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Αυτό ήταν το επιχείρημα που τελικά μας επέτρεψε να επιβάλλουμε την άποψή μας επ' αυτού. Τα καταφέραμε ενώ υπήρχε μεγάλη πίεση χρόνου όπως όλοι γνωρίζετε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Γιατί έτσι θα ξεκινήσει το EDIDP την 1η Πρώτου 19. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Θα ψηφίσουμε σε δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους της ΣΕΝΤΕ και στις άλλες επιτροπές που συμμετείχαν για τη συνεργασία τους. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την γνωμοδότηση ΑΦΕΤ συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του EDIDP μέσω της ουσιώδους ε, συμβολής του τριμερούς διαλόγου. Αυτό θα μπορούσε να είναι έμπνευση και για τις επόμενες προτάσεις της Επιτροπής για την υπόλοιπη διάρκεια του επομένου πολιετούς πλαισίου. Εν συντομία αυτά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ πλήρη παρουσίαση. Έχουμε κάποιο χρόνο για συζήτηση, περιορισμένο βέβαια, αλλά έχουμε. Κύριος Κέλαμ, θέλει το λόγο κύριε Μόντι. Όχι, ναι. Κύριε Μόντι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Είπατε ότι το 60% προέρχεται από υπάρχοντα προγράμματα. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ποια είναι αυτά. Uh, Κύριε Κέλλαμ θέλετε το λόγο? Όχι. Κύριε Βαλέρο. Κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, αν θέλετε. Πρώτον, δεν ξέρω αν είναι ε, υπόθεση εργασίας ή πραγματικότητα, αλλά φαίνεται ότι διοχετεύονται ποσά σε πολύ ισχυρέ αμυντικέ βιομηχανίε στην Ευρώπη ε, που δεν χρειάζονται στήριξη. Γιατί είναι ήδη ισχυρές επιχειρήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται να τις ε, στηρίξουμε με πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, που το είχα γραμμένο, δεν μπορώ να το βρω. τα έχω γραμμένα στα γερμανικά και δεν βγάζω τι έχω γράψει. Yeah, the other one, yeah, I'm sorry. The other, the other question I have is... Ναι, το θυμήθηκα. Τι, άλλους, τι περιορισμούς έχουμε, θέτουμε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα όπλα, αυτός ο εξοπλισμός δεν θα καταλήξει σε χώρες όπως η Εμένη, η Συρία ε, σε εμπόλεμες ζώνες ε, ε, και για να μην συνεισφέρουμε στην επιμήκυνση και την παράταση αυτών των σειράξεων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να κάνω μία ερώτηση. Για αυτό το 60%, 60-40. Έχουμε μία γενική ιδέα για το πού ενδεχομένως έχουμε ε, διαθέσιμα κονδύλια. Το καταλαβαίνω, μα μιλήσατε για 60-40%. Αλλά αυτό το 60, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, πού θα προέρχονται αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, το γνωρίζουμε ήδη ή θα αποφασιστεί αργότερα. Νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω το λόγο, κύριε Πάσκο. Κυρία Μούντι. Το Συμβούλιο και γενικότερο τεμερής διάλογος ε, ανέφερε, αποφάσισε ότι 116,1 εκατομμύρια από το CEF, 3,9 από το ΕΓΝΟΣ, 104,1 από το Γαλιλαίο, 12 από το Κοπέρνικος 63,9 εκατομμύρια από το ITER. Αυτές, αυτά θα είναι, αυτές είναι οι γραμμές από τις οποίες θα πάρουμε χρήματα. Η ανάλυση έγινε από την Κομισιόν και μας ε, βεβαίωσε η Κομισιόν ότι δεν θα επηρεάσει την ε, εξέλιξη των άλλων προγραμμάτων και μας, γιατί, ε, το, γιατί ανησυχούσαμε. Μα είπε η Κομισιόν ότι αυτά τα χρήματα είναι διαθέσιμα, δεν θα επηρεάσει αυτή η μεταφορά τη λειτουργία των άλλων προγραμμάτων. Το Κοπέρνικος 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια από το Κοπέρνικο. 63,9. 104 εκατομμύρια από το Γαλιλαίο. Αυτά είναι τα νούμερα. Πάντως η Κομισιόν μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει επίδραση στην λειτουργία και την εξέλιξη των προγραμμάτων. Και θα ήταν παράλογο να πάρουμε χρήματα από άλλα προγράμματα, να τα ε, φέρουμε εδώ και να δημιουργήσουμε προβλήματα αλλού, δηλαδή να μετακινήσουμε το πρόβλημα σε άλλα προγράμματα. Για τη δεύτερη ερώτηση, για τις πολύ ισχυρές εταιρείε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι μεγάλες εταιρείε ε, δεν θα χρηματοδοτηθούν επειδή έχουν δικά τους λεφτά. Δεν μπορούμε. Οι συνθήκες, οι όροι είναι ίδιοι για όλους. Αυτό όμως που θέλουμε να εξασφαλίσουμε και ακριβώς επειδή γνωρίζαμε πώς θα προσπαθήσουν να συμμετάσχουν μεγάλες εταιρείε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν επίσης επίσης όρης. Οπότε η φιλοσοφία δεν ήταν να αποφύγουμε τη συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτές είναι που ε, αποτελούν την ουσία της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Αυτές έχουν την υποδομή και τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για να καινοτομήσουν. Οπότε θα ήταν σαν να δέναμε το ένα χέρι μας πίσω από την πλάτη μας, αν τους απαγορεύαμε να συμμετάσχουν. Όμως προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πιο μικρές εταιρείε και οι εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης ε, θα ε, συμμετάσχουν επίσης όλοι στο πρόγραμμα. Με τις εξαγωγές τώρα. Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα για την ανάπτυξη συγκεκριμένου εξοπλισμού και μετά να απαγορεύσουμε τις εξαγωγές. Υπάρχουν και θέματα τεχνίας. Αν θέλαμε να ελέγξουμε τις εξηγήσει, θα έπρεπε να το δούμε πιο γενικά. Ε, έχουμε άλλα εργαλεία τα οποία ε, προλαμβάνουν την ε, εξαγωγή σε περιοχές στις οποίες δεν θέλουμε. Μετά τα δύο χρόνια άλλωστε του προγράμματος θα δούμε, κάνουμε και ένα απολογισμό για να δούμε πώς λειτουργεί. Τώρα, για τους τομείς ε, θα καλύπτονται καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες που στην προετοιμασία, προστασία, ανάπτυξη και ε, ε, στην ε, διαχείριση της πληροφορίας, συστήματα αναγνώρισης, κυβερνοάμυνα και κυβερνοασφάλεια, αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά είναι οι τομείς στους οποίους θα δώσουμε έμφαση. Αν είμαστε πολύ περιοριστικοί, δυσκολεύουμε την καινοτομία. Οπότε θελήσαμε να είμαστε αρκετά ευρείς χωρίς όμως να είμαστε και να, χωρίς όμως να ανοίξουμε υπερβολικά το πεδίο. Ο Γκάλερ θέλει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να μιλήσω στην ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Χωρώνα και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια. Γι' αυτό ο καθυστέρησα. Ε, με χαρά βλέπουμε να υιοθετείται αυτή η έκθεση από την Επιτροπή. Τρέμε μάλιστα με ισχυρή πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Νομίζω το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Να σας θυμίσω ότι η αμυντική βιομηχανία έχει εκφράσει το φόβο ένα φόβο που έχει σχέση με την έρευνα και με την ανάπτυξη βέβαια ε, για το γεγονός ότι ο πελάτης είναι το κράτος και όταν αυτά τα προγράμματα γίνονται σε εθνικό επίπεδο, το κόστος της αμυντικής βιομηχανίας, τα κόστη της αμυντικής βιομηχανίας είναι πάνω από 100%. Οι ίδιοι λένε πάνω από 125%. Η επιστροφές ε, φοβούνται ότι δεν θα καλύπτουν όλο το κόστος της επιχείρησης. Εδώ έχουμε ένα πραγματικό ερωτηματικό. Η, η, η αμυντική βιομηχανία φοβάται ότι θα πρέπει να βάλει πιο πολλά χρήματα από ό,τι θα πάρει από το πρόγραμμα. Το άλλο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξή. Το αποτέλεσμα θα πρέπει τελικά να είναι χρήσιμο για το στρατό μα. Ε, δεν θα πρέπει απλώ να εξυπηρετήσουμε την αμυντική βιομηχανία. Το στρατό μα, του στρατούς μας θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Αυτοί θα πρέπει να ικανοποιηθούν από το αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα λοιπόν θα πρέπει να βοηθάει με αυτό τρόπο, όχι θεωρητικά μόνο, τα στρατεύματά μας. Τα στρατεύματά μας θα πρέπει να δηλώσουν τι χρειάζονται και η αμυντική βιομηχανία να τα παράσχει. Κύριε Πάσκου, συμφωνώ απόλυτα το γεγονός ότι ε, στην πράξη πελάτης είναι το κράτος γιατί την εθνική αρμοδιότητα η άμυνα ε, είναι ένας κίνδυνος. Δεν περιμένουμε ότι οι εταιρείε θα κάνουν βασική έρευνα. Ε, εφαρμοσμένη έρευνα θα κάνουν. Γιατί θα πρέπει να παρέχουν αυτά που χρειάζεται ο στρατός. Πάντως καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών και το 25% των έμεσων δαπανών. Αυτή είναι η διάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ε, είμαστε ευγνώμονες στον κύριο Πάσκο για τις προσπάθειές του και για τις παρουσιάσεις που μας έκανε τρεις-τέσσερις φορές. Μας παρουσίασε τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Προλαβαίνουμε να ψηφίσουμε το θέμα στην επόμενη ολομελία μας. Θέλετε να σχολιάσετε? Όχι, σας ευχαριστώ που με ευχαριστείτε, τίποτα άλλο. Ωραία. Μπορούμε απλώς λοιπόν να αλλάξουμε τους συμμετέχοντες στο Προεδρείο για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Παρακαλώ να μείνετε στην αίθουσα. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Επόμενο σημείο στην εμερήσια διάταξη, εφαρμογή του προγράμματος δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Θαλάσσιας Ασφάλειας. Είναι χαρά μου να υποδεχτώ τους συμμετέχοντες ε, στο πάνελ. Πρώτα απ' όλα την πρέσβυρα Γεωργιάνα Καρατζόβα, εκπρόσωπο της ε, τρέχουσας βουλγαρικής προεδρίας, διότι σε αυτό το εξάμεινο βρισκόμαστε στην ε, βουλγαρική προεδρία Εδώ έχουμε τον κύριο Μπένχαρντ Φρίς της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ υπεύθυνο για θέματα θαλάσσιας ε, ε, και γαλάζιας οικονομίας. Μετά ο πρέσβης Χαζίνσκι, διευθυντής στον ΙΕΣ, και μετά ο γνωστός και πολύ προσκληθής στην αίθουσα αυτή και σήμερα ο πρέσβης Ζόρζε Ντόμεκ διευθυντής για τα θέματα ε, μάλλον στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ξεκινάμε με την πρέσβηρα Καρατζόβα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μας υποδέχεστε, ε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. προσκεκλημένοι της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ, θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας την εκτίμησή μου για την συμπερίληψη του θέματος της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής ε, Στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας και του σχετικού προγράμματος δράσης στην και κατέξη της ε, ΣΕΝΤΕ. Η αναθεώρηση της, ε, του προγράμματος δράσης για στρατηγική και η έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την αναθεώρηση αυτή αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο ε, που απασχόλησε τη Βουλγαρική Προεδρία στο πεδίο των των, πραγμα, των υποθέσεων της θάλασσας. Ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία με την ε, Προεδρία και την ΕΙΕΔ, τις ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική ε, Διεύθυνση, τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Έτσι κατέστη δυνατή αυτή η προσπάθεια. Ήθελα να πω ότι στο πνεύμα διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή σας είναι όντως απαραίτητη. Για τη διαδικασία και τα βήματα για το μέλλον. η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής θαλάσσιας, Στατικής Θαλάσσιας Ασφάλειας είχε να κάνει με τον ρόλο που θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνούς παράγοντα στα θέματα αυτά. Η διεύρυνση της στρατηγικής αυτής έχει σχέση με την ε, παγκόσμια στρατηγική και τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των άλλων συμβουλίων. Το 2014 το πρόγραμμα δράσης, το αρχικό πρόγραμμα δράσης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας συνδυάσαμε εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ενωσιακής θαλάσσιας ασφάλειας. Η αναθεώρηση του προγράμματος δράσης σκοπό έχει να προχωρήσει στην καλύτερη υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ε, την αναθεωρημένη ε, στρατηγική εσωτερική ασφάλεια 2015-2020 και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου για την Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Ασφάλεια χρήζουν επικαιροποίησης και αναθεώρησης. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης βασίζεται στις αρχές της στατικής που έχουν συμφωνηθεί. Την διατομεακή προσέγγιση, την εξωτερική δράση, την ευαισθητοποίηση, εποπτεία και ε, πληροφόρηση, την ανάπτυξη δυνατοτήτων, τη διαχείριση κινδύνου, την προστασία κρίσιμων ε, υποδομών και απόκριση τη κρίση, την έρευνα για την ασφάλεια και καινοτομία, την εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του σχετικού προγράμματο δράση, λοιπόν, και το αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης αποτέλεσαν παράρτημα στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, όπω τα συμφώνησα η ομάδα φίλων τη Προεδρία στι 25 Μαΐου. Τη συμφωνία την επιβεβαίωσε το Κορεπέρ στι 13 Ιουνίου και τα δύο έγγραφα θα πρέπει να εγκριθούν από κοινού στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 26 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας οργανώθηκαν έξι συνεδριάσεις ε, της ομάδας φίλων της Προεδρίας και εξετάστηκε ένα non-paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της είπα της εκπροσώπου για την αναθεώρηση, πράγμα που κατέλησε βάση των διαπραγματεύσεων. Στη βάση αυτών των συζητήσεων η Προεδρία ε, εκπώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδας φίλων της Προεδρίας το Μάιο έγινε, επιτελέστηκε σημαντική πρόοδος για να επιτευχθεί ο στόχος της Βουλγαρικής Προεδρίας. Επιπλέον, η αναθεώρηση τη σχετική στρατηγική και του προγράμματο δράση τη συμπεριλήφθηκε στην ατζέντα του πίεση στις 8 Μαΐου. Εκεί σημειώθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για το πρόγραμμα δράσης και επιβεβαιώθηκε η σημασία του προγράμματος δράσης για να ε, ε, υλοποιηθούν οι δράσεις της ε, παγκόσμιας στρατηγικής. Η εθελοντές πρωταθλητές όπως ε, ονομάστηκαν είναι από τους σημαντικούς ε, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δράσης αυτό και όλα αυτά περιλαμβάνονται και στα ενημερωτικά σημειώματα της ε, Προεδρίας σε έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένε προτάσει. Τώρα, διαφορέ μεταξύ του προγράμματο το 2014 και το 2018. Το αναθεωρημένο, το καινούριο δηλαδή πρόγραμμα δράση έχει μια ανανεωμένη ε, δομή με το τμήμα Α για τα οριζόντια ζητήματα και το τμήμα Β για τις περιφερειακές υποθέσει ώστε να ασχοληθεί με μια περιφερειακή προσέγγιση στι ε, θαλάσσιε λεκάνε και του τέσσερι ωκεανού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα δομή και η προσέγγιση έγιναν δεκτά με πολύ θετικό τρόπο από τα κράτη-μέλη και θα συνδυαστούν με άλλε εξελίξει στι ε, πολιτικέ και περιφερειακέ στρατηγικέ. Επίσης, το αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης ευθυγραμμίζεται το αρχικό πρόγραμμα δράσης το 2014 ως προς την έμφαση στην ε, ε, συνεργασία ε, στον τομέα των πολιτικών και στρατιωτικών υποθέσεων, την διεθνή συνεργασία, την κατανομή πληροφοριών, την ανάπτυξη δυνατοτήτων, και τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, ιδίως την παγκόσμια στρατηγική και το τι συμβαίνει στη θάλασσα με τη μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο. οι τομεακές και περιφερειακές ε, στρατηγικές ε, που ε, εφαρμόζονται στις θαλάσσιες λεκάνες και τους κοινούς θαλάσσιους χώρους στον ευρύτερο τομέα των θαλασσών παγκοσμίω ε, είναι, είναι στοιχεία που ανταποκρίνονται πλέον σε συγκεκριμένε δράσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώ. Το ίδιο και με την ΚΑΡ, την ΠΕΣΚΟ και την ΕΝΤΑΠ ε, που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής. Όπως θα ξέρετε, Όλα αυτά θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν και οι πολιτικές δυνατότητες, όπως θα αποφασιστεί αργότερα φέτος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η πρόταση που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο για την υλοποίηση της κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και των σχετικών συμπερασμάτων του Συμβουλίου. και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες των κρατών μελών, των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών της για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις προς την ασφάλεια ε, και οι, κυβερν... οι κυβερνοαπειλές, οι και τρομοκρατικές απειλές και απειλές από χημικά και βιολογικά όπλα, ώστε να έχουμε καλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα. Ίσως μόνο το follow-up τώρα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δράσης έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα εξελίξει ζωντανό κείμενο το οποίο θα ε, υποβάλλεται σε τακτική αναθεώρηση βάσει των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης και σε επικαιροποίησης. Θα είναι επίσης ένα διαρκές εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων από τα κάτι μέλη, τα οποία θα ενημερώνονται και θα ενημερώνουν και τους σχετικούς ε, συμμετέχοντες στην όλη στρατηγική. Το ίδιο και τα σώματα καθώς και οι ομάδες εργασίας που αποτελούνται από πυροχνόμονες και που ασχολούνται με την πρόοδο και την υλοποίηση του προγράμματος. Director... Ευχαριστώ. Και τώρα από την DGMAR ο Διευθυντής κύριος Μπερνά Φρίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμα μέλη. Καλημέρα σας. Με χαρά είμαι σε αυτή την αίθουσα και είναι κατάλληλη στιγμή για να σας ενημερώσω για την εργασία που κάνει η υπηρεσία μου για το σχέδιο δράσης του EU MSS. Τη στρατηγική μας για την θαλάσσια ασφάλεια, δηλαδή της Ένωσης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και ελπίζω ότι θα είναι υποφελής αμοιβαία συζήτηση. Θέλουμε να έχουμε μια ακόμη ευρύτερη προσέγγιση έναντι των ωκεανών που είναι θεμελιώδους σημασία από οικονομική, περιβαλλοντική αλλά και από πλευρά ασφάλειας. Το 90% του εμπορίου είναι θαλάσσιο. 50% του πλησμού της Ένωσης ζει σε παράκτης περιοχές. Δηλαδή λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από την παραλία. 400 εκατομμύρια επιβάτες περνάνε από τα λιμάνια μας κάθε χρόνο. Άρα τίθεται ένα ακόμη ευρύτερο πλαίσιο. Η Ένωση έχει και μια πολιτική για την διακυβέρνηση των ωκεανών για να διαχειριστούμε τους ε, ωκεανούς μας με υπεύθυνο τρόπο. Η EU MSS άρχισε να λειτουργεί το 2014. Δεν θα επαναλάβω τη διαδικασία εκπόνησής της γιατί την έκανε η κυρία Πρέσβης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προποθέσει που υπήρχαν το 2014 εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες προκλήσεις, σε νέες επίγουσες καταστάσεις. Για το 2014 μέχρι 2018 έχουν περάσει 4 χρόνια. Έχει αλλάξει η προσέγγιση από πλευρά των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην θαλάσσια ασφάλεια. Έχει αυξηθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων, μεταξύ διαφόρων φορέων, οργανισμών, στρατιωτικών και μη. Ίσως στο παρελθόν όλα αυτά να μην ήσαν προφανή. Αυτό νομίζω ότι είναι επίτευγμα του σχεδίου δράσης και πρέπει να πάμε και πιο μακριά. Όπως σας είπα, τη διαδικασία δεν θα την επαναλάβω. Ποια είναι τα σημαντικά νέα στοιχεία και οι νέες προτεραιότητες για αυτήν την αναθεώρηση με βάση των κατευθυντηρίων αρχών του σχεδίου δράσης του 2014 Το εξακολουθούν να ισχύουν <clears throat> και πρέπει να ε, υλοποιηθούν. Με χαρά σημειώνουμε ότι αυτή η αναθεώρηση θέλει να αυξηθεί η περιφερειακή συνεργασία. Ναι μεν Ευρώπη, αλλά και περιφέρειες. Μεσόγειος για παράδειγμα. Η αρχική πολιτική όθηση για να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα δράση ήταν η μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο με όλα τα ανθρωπιστικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας που θέτει. Στη Μεσόγειο ακριβώς επιδιώκουμε μια ευρύτερη συνεργασία. Για παράδειγμα, έχουμε την ε, θαλάσσια στρατηγική για τη Δυτική Μεσόγειο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ πέντε αφρικανικών και τριών ευρωπαϊκών χωρών με ανταλλαγή προφοριών Όποιο ακούει τα νέα διαπιστώνει βέβαια ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές προκλήσεις στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα επίσης Πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην περιοχή. Για βέλτιστη, για παράδειγμα, αντιμετώπιση του προβλήματος των χημικών αλλά και άλλων όπλων που τα ρίχνουν στη θάλασσα και για άλλα προβλήματα και δημιουργούν διάφορα προβλήματα βέβαια στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην αλία στον Ατλαντικό που είναι επίσης άλλη ζωτική σημασία θαλάσσια έκταση πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παράνομες ναυτικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή όλων των φορέων όπως το κέντρο για παράδειγμα για την ανάλυση και τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπιστεί η μεταφορά ναρκωτικών πρέπει να υπάρξει περισσότερο πνεύμα συνεργασία. Βεβαίω ε, όλοι έχουμε συνέστηση των δυσκολιών δεν χρειάζεται να τι εξηγήσω αλλά αν είμαστε ρεαλιστέ υπάρχουν δυνατότητε να δημιουργηθούν μορφές συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι κοινέ προκλήσεις. Η περιφερειακή προσέγγιση είναι σημαντική και θα εξακολουθήσει να είναι και να γίνεται πιο σημαντική. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων. Αυτός είναι ένας από τους κύριους ε, στόχους του υπάρχοντος ε, προγράμματος δράσης Πρέπει να υπάρξουν κοινέ πρωτοβουλίε για την ε, ανάπτυξη δυναμικού και περισσότερη συνεργασία γενικότερα σε επίπεδο ένωσης. Και η νομοθεσία και οι πόροι που εγκρίνεται ως Κοινοβούλιο μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των τριών φορέων που ασχολούνται με τη θάλασσα, την Frontex, τον Οργανισμό για τον Έλεγχο της Αλίας και τον Οργανισμό για τη Θαλάσσια Ασφάλεια της Λισαβόνας. Αυτή η συνεργασία είναι προστιθέμενη αξία. Αυτή η συνεργασία έχει επεκταθεί σήμερα και σε πάνω από 300 ε, πολιτικές ε, και άλλες υπηρεσίες ακτοφυλακής των κρατών μελών που συνεργάζονται για την ασφάλεια, για την έρευνα και διάσωση, για τον έλεγχο των συνόρων, τον έλεγχο των αλληλευμάτων, τα τελωνία, την εφαρμογή του νόμου, την προστασία του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία δηλαδή που σας δίνει ένα drone ή οποιαδήποτε δραστηριότητα επιτήρησης από ένα φορέα μπορούν να ε, δοθούν και σε άλλους για παράδειγμα, ε, διάφορα αεροσκάφη που επιτηρεί την ε, αλληλευτική δραστηριότητα εντοπίζει ένα σκάφος ε, που κινδυνεύει να βυθιστεί με μετανάστες και ενημερώνει τους άλλους φορείς. Εδώ η συνεργασία δουλεύει πολύ καλά, αλλά πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Άλλο τομέα συνεργασία. Επίση ζωτικό. Ενταλλαγή πληροφορίε για την αυτιλία. Έχουμε λειτουργικά συστήματα που λειτουργούν και μας δίνουν μια ε, ενοποιημένη εικόνα για την ναυτιλία. Κυρίως ε, συντονίζει αυτή τη δραστηριότητα ε, ο ΕΜΣΑ στη Λισαβόνα. Μπορεί όμως να βελτιωθεί αυτή η δραστηριότητα και θέλουμε να ξεκινήσει και το ΣΥΖΑ, το κοινό περιβάλλον για την ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, το αναθερημένο πρόγραμμα δράσης θα εξετάσει και τις αναδυόμενες απειλές, για παράδειγμα κυβερνοαπειλές, υβριδικές, γιατί η αυτοματοποίηση και η χρήση πληροφορικής επεκτείνεται. Για παράδειγμα υπάρχουν, ε, αρχίζουν να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα αυτόματα πλοία. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι ασφαλής μπορούν να προκύψουν. Πρέπει να προστατεύσουμε βέβαια και τις ζωτικές υποδομές, για παράδειγμα, τις λιμενικές. Και αυτές είναι βασικές προτεραιότητες. Επίσης, πρέπει να προστατεύσουμε και τους επιβάτες ε, στις θαλάσσιες μεταφορές. Βεβαίως πρέπει να διατηρούνται ανοιχτές ε, <coughs> συγγνώμη οι επικοινωνίες μας επίσης περνάνε από υποθαλάσσια καλώδια πρέπει να τα προστατεύσουμε και αυτά και χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση κάθε τομέας που μπορεί να ε, κινδυνεύει η ασφάλειά του και βέβαια πρέπει να προβλέψουμε και τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Ένα πρόγραμμα δράση που είναι ανοιχτό προ το μέλλον είναι η σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ του συναδέλφου για τη συνεργασία <clears throat> και προσβλέπω στην υιοθέτηση από το Συμβούλιο τη Νέα ε, Προσέγγιση, το νέο πρόγραμμα δράση. Και τώρα ο κύριο Παύλ Χερτουίνσκι του EEAS, Αρμόδιο για την πολιτική ασφάλεια. και την πρόληψη συγκρούσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και την Πρόεδρο την κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε για ένα τόσο επίκαιρο ζήτημα ε, εν ώψη της ε, ε, ε του ε, από το Συμβούλιο ε, της, ε, του καινούριου προγράμματος θαλάσσιας ασφάλειας. Η πρέσβης κυρία Καντήροβα ήταν πολύ μετριόφρον παρουσιάζοντάς μας τα διάφορα στάδια τα οποία χρειάστηκε να περάσει το Συμβούλιο για την υιοθέτηση αυτού του εγγράφου. Για μας η βουλγαρική Προεδρία τα κατάφερε πολύ γρήγορα. Έχουμε κάνει σημαντικότατη πρόοδο σε τους τρεις τελευταίους μήνες. Και αυτό χάρη και στην υποστήριξη όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και της πολύ καλής συνεργασίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Από τη δική μας οπτική γωνία, το καινούριο πρόγραμμα δράσης είναι βασικό στοιχείο για την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊ... Παγκόσμιας Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι περιμένουμε από αυτό το πρόγραμμα δράσης. Από την ε, πλευρά της εξωτερικής δράσης στόχος είναι η, η θαλάσσια στρατηγική να εναρμονιστεί με την παγκόσμια στρατηγική και να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, παγκόσμιος πάροχος ε, ασφάλειας στη θάλασσα. Οι βασικές αρχές ε, της ε, θαλάσσιας ασφάλειας παραμένουν. Για παράδειγμα, η καθολικότητα της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ και ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα όμως, το καινούριο πρόγραμμα δράση θέτει την έμφαση στην ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία και σε διεθνείς πτυχές η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω περιφερειακών απαντήσεων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του καινούργιου γράφου. Τοπικές δράσεις που θα απαντούν σε παγκόσμιες προκλήσεις. Ε, αυτό αφορά ε, και το κέρας Αφρικής και την Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και τη Μεσόγειο ε, που είναι το κατόφλι μας. Αυτή η προσέγγιση είναι καινούργια και γι' αυτό λόγο εν συντομία θα ήθελα να σας παρουσιάσω ορισμένες από τις βασικές προτάσεις. Συνεργασία στη θάλασσα είναι μία από τις πιο ορατές πτυχές της ασφάλειας θάλασσα. Στη Μεσόγειο η συνεργασία με το ΝΑΤΟ σε επιχειρηματικό επίπεδο ε, μέσω της ε, επιχείρησης Σοφία και της Sea Guardian ε, είναι βασικά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και για να σώσουμε ζωές στη θάλασσα. Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι βασικός ε, παράγοντας του, της δράσης, του προγράμματος δράσης και θα πρέπει να συνεισφέρει στην ε, υλοποίηση του θαλάσσιου πυλώνα της συνεργασίας που φασίστηκε στην Βαρσοβία και θα μπορούσε μάλιστα να διευρυνθεί και σε άλλες περιοχές κοντά μας, ε, όπως για παράδειγμα την Μαύρη Θάλασσα. Πολύ δε περισσότερο που η περιοχή αυτή ε, στατιωτικοποιείται όλο και περισσότερο και χτίζεται και η γέφυρα που θα ενώνει, η γέφυρα που θα ενώνει ε, την Κρυμαία με την Ρωσία. Ένα άλλο σημείο για τη Μεσόγειο είναι η βελτίωση της συνεργασίας και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ε, αποστολές ε, ε της ε, της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και, τον, και του πυλώνα της ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ε, συγγνώμη, της, του Τζάι η, πάντοτε είχαμε συνεργασία ε, μεταξύ ε, αυτών των δύο, αλλά ήταν, ε, είχε πολλά προβλήματα αυτή η συνεργασία και θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Ε, ξεκινάμε ένα πολιτικό πρόγραμμα που θα ενώνει τις υπηρεσίες του, του πυλώνα Τζάι με τις αποστολές μας που έχουν σχέση με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας χρειάζεται. Ε, αυτά τα δύο, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικέ υποθέσει να και, η, ε, και η ασφάλεια και η άμυνα να ενωθούν, ε, να συνεργαστούν. Μετά, ε, ο Ινδικός ωκεανός είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας και θα πρέπει να παραμείνουμε σημαντικοί παίχτες. Γι' αυτό το λόγο, η οι χώρες ε, ΚΟΑΖΙ που είναι ε, αυτές που συνδέονται με τις... Ε, είναι 26 χώρες που, που σχετίζονται με τον Ινδικό ωκεανό συνεργάζονται και τα κράτη-μέλη επιθυμούν μια στρατηγία τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Να σας πω πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από το κέρας Αφρικής ό,τι αφορά την πολιτική μας θάλασσα. Σήμερα αυτή η περιοχή δεν είναι αποκλεισμένη για μας. Ε, οι πειρατικές επιθέσεις έχουν μειωθεί πολύ σε μεγάλο βαθμό χάρη ε, στην επιχείρηση Αταλάντα και την γενικότερη διεθνή παρουσιακή. Έχουμε όμως και άλλες προσπάθειες όπως η των βέλτιστων πρακτικών τις οποίες ε, ακολουθεί ο κλάδος. Ε, τον Ιούνιο θα υιοθετήσουμε ένα καινούριο ε, σετ ε, συμπερασμάτων για την Ερυθρά Θάλασσα και το κέρας Αφρικής. Εμείς στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης προσπαθούμε να επωφεληθούμε από την εμπειρία μας εναντίον της πειρατείας εκεί για να αντιμετωπίσουμε και άλλου τύπου εγκλήματα στον Ινδικό ωκεανό, στην, από την ε, Θάλασσα μέχρι την Ιεμένη και τον πορθμό του, της Μάλακα. Ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε επίση τα συμπέρασματά μας και στον κόλπο της Γουινέας, ε, όπου υποστηρίζουμε τη διαδικασία της Γιαουντέ και την δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη ε, ε μιας διαδικασίας καλύτερης αντίληψης της κατάστασης. Τέλος, να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία με τον ΟΗΕ έχει ενισχυθεί με το νέο, ενισχύεται μάλλον με το νέο πρόγραμμα δράσης. Θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο για το μέλλον των ωκεανών, λαμβάνοντα υπόψη ότι η στρατηγική ε, εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ, και ΝΑΤΟ, συγγνώμη, ε, και, και ΟΗΕ, ε, περιλαμβάνει πλέον και τους ωκεανούς. το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ είναι δύο από τους ε, βασικούς εταίρους μας ε, στη θάλασσα, η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τον ΑΣΕΑΝ, καθώς επίσης και με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, παραμένει επίσης σημαντική. Το κείμενο του προγράμματος δράσης ε, προβλέπει ότι το πρόγραμμα δράσης θα αναθεωρείται με βάση εκθέσεις που θα γίνονται τακτικά. Ε, το ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να ε, βελτιωθεί η ε, συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο, σε συνεργασία με την Βουλγαρική Προεδρία, ξεκινάμε κάποια βήματα για την ανάπτυξη, την προετοιμασία υλικού, επικοινωνιακού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί με την υιοθέτηση του προγράμματο δράση, για παράδειγμα, για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και για το κέρα τη Αφρική δύο μέρες πριν την υιοθέτηση αυτού του εγγράφου μπορούμε να είμαστε ε, χαρούμενοι και περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει που όμως αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Ε, θα χρειαστεί και άλλες δράσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο πρέσβης Χόρχε Ντόμεκ υποδιευθυντή στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα δράση για την θαλάσσια στατική ασφάλεια που προβλέπεται να εγκριθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου την εβδομάδα είναι έγκαιρη και σκόπιμη. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη διάσταση τη άμυνα αυτό το πρόγραμμα δράση. Έχουμε νέε εξελίξει για τι πρωτοβουλίε άμυνα και ασφάλεια ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω την, την και προκειμένου να υλοποιηθεί νέα παγκόσμια στρατηγική καθώς και ενισχυμένη συνεργασία με το ΝΑΤΟ όπως είπε και ο πρέσβης. Θα ήθελα να τονίσω ότι το να έχουμε αμοιβαίως ενισχυόμενες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και την ε, ε, άμυνα και σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι στόχος του αναθεωρημένου ε, προγράμματος δράσης και συνιστόσα τη παγκόσμια στρατηγική. Αυτό και για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που χρειάζονται τα τη στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων. Όπως ξέρετε, είναι βασική αρμοδιότητα του Οργανισμού για την Άμυνα να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μέσω της συνεργασίας. Ο οργανισμός μας ήδη διδραματίζει κεντρικό ρόλο σε όλες αυτές τις πρόσφατες εξέλιξεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Προκειμένου να το πράξουμε αυτό, προσαρμοζόμαστε στο νέο, ε, στις νέες με την μακροπρόθεσμη αναθεώρηση όπως την ανέκριναν οι Υπουργοί πέρσι τον Μάιο. Επίσης, οι αρμοδίτες μας προβλέπουν ρόλο διεπαφής διαμεσολαβητή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων, καθώς και των μεγαλύτερων οργανισμών μας, ώστε οι ένοπλε δυνάμει μα να μην έχουν αρνητικέ συνέπειε να μην περιοριστούν στη δράση του. Να τονίσω ότι ο ρόλο διεπαφή, όπω έχει ονομαστεί, έχει σημαντική βαρύτητα στον τομέα της θάλασσας. Μια από τι βασικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα είναι η διατομεακή προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει και πολιτικέ και στρατιωτικέ πτυχέ και παράγοντε ζωτική σημασία για να μπορέσουμε αποτελεσματικώ να αντιμετωπίσουμε απειλέ στη θαλάσσια ασφάλεια. Έτσι, η βασική συνεισφορά του οργανισμού μας στην υλοποίηση του πρόγραμματος δράσης θα προκύπτει από τη βασική μας εντολή σε τομείς όπως η ανάπτυξη δυνατοτήτων, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, καθώς και η έρευνα και η καινοτομία. Η σε εξέλιξη αναθεώρηση του προγράμματο δράση για την ανάπτυξη δυνατοτήτων που τώρα επικεντρώνεται περισσότερο στα αποτελέσματα, προχωρεί και επικεντρώνεται ακριβώ στι δυνατότητε και το τι επιδιώκουν τα κράτη-μέλη και στον τομέα τη θάλασσα. Οι νέε προτεραιότητε θα συμφωνηθούν στο τέλο του μήνα από αυτήν την οπτική γωνία η θεώρηση της Ευρωπαϊκής ε, Στατικής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια και το πρόγραμμα δράσης της είναι επίκαιρη, διότι για την υλοποίηση του πρόγραμματος δράσης πρέπει να προχωρήσουν ε, οι δυνατότητές μας και η ανάπτυξή τους ε, στην θαλάσσια ασφάλεια και βάσει των προτεραιοτήτων της ΚΕΠΑ, ιδίως για τις θαλάσσιες δυνατότητες που μπορεί να έχουν πολλαπλή χρήση. Ένα σαφέ παράδειγμα τέτοιων δυνατοτήτων που ανέπτυξε ο οργανισμός είναι το πρόγραμμα θαλάσσιας παρακολούθησης μάσου το οποίο συνδυάζει 18 ε, ναυτικές δυνάμεις, 18 στόλους με σκοπό να έχουμε μια συνολική εικόνα για τα πράγματα στη θάλασσα και την ανταλλαγή επιχειρησιακών ε, πληροφοριών και υπηρεσιών στη θάλασσα, όπως τη θέση των σκαφών, τα ίχνη, ε, τα τσάτ και τα μηνύματα ή τις εικόνες. Ε, το Μασούρ ήδη χρησιμοποιείται στη, και χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση Σόφια και θα ενισχυθεί με, νέα τεχνολογικά μέσα ε, είναι το μόνο στρατιωτικό εργαλείο του είδους του και μπορεί να δώσει μια ενιαία στρατιωτική εικόνα στο περιβάλλον των κοινών πληροφοριών για τις θαλάσσιες τεχνικές ε, πληροφορίες. Η σημασία του Μασούρ ε, ε, τονίστηκε και στα συμπράγματα του Συμβουλίου πέρσι και είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί και στο νέο πρόγραμμα δράσης. Οι δυνατότητε αυτές θα εξυπηρετήσουν και τον πρωταρχικό στρατιωτικό μας σκοπό, αλλά θα συμβάλλουν και στι αρμοδιότητε προστασία των πολιτών, τη πολιτική προστασία, που είναι βασικό στόχο του προγραμματός δράσης. Μια, ένας άλλος τομέας προτεραιότητας για τον οργανισμό μας είναι η έρευνα, η πρωτογενής έρευνα και το σχετικό εργαλείο ιεράρχησης ε, επιτρέπει στην συνολικότερη ατζέντα για την έρευνα, την όσρα, να συνδυαστούν με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα προγράμματα δράσης των κατώμελών. Βάσει της πείρας μας ως τώρα, ο συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων του οργανισμού καθώς και των προγραμμάτων χρηματοδότησης ε, και έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα λόγου χάρη κρίσης είναι ένας ελπιδοφόρος ορίζοντας που ήδη δίνει σημαντικά αποτελέσματα όπως με τα επιτεύγματά μας το σχετικό ε, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα Horizon 2020 καθώς και τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα και πράγματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διπλή χρήση. Για να τονίσουμε περισσότερες σχέσεις συνεργασίας, εμπειρογνώμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΕΔ και τον Οργανισμό Άμυνας, καθώς και τα κάτι μέλη και τις εταιρείε, έχουν συνεργαστεί για να δημιουργηθεί μια διαταμιακή ατζέντα για την θαλάσσια ασφάλεια. Ένα από τα συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα που θα επιδιωχθούν στην υλοποίηση της ε, στρατηγικής της θαλάσσιας ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα αυτό που μας απασχολεί είναι η υλοποίηση όπως ε, ε, αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα δράσης όπως αναθεωρήθηκε. Στον τομέα της ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης τώρα, εδώ θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια τομεακή προσέγγιση και κουλτούρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, η δουλειά μας εδώ σκοπό έχει να προβλέψει κύκλους κοινή εκπαίδευση για θαλάσσια θέματα και την ευαισθητοποίηση στα θέματα της θάλασσας. Για όλες αυτές τις προσπάθειές μας, η έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και ε, κατάρτιση, ο εντοπισμός και η διαχείριση κινδύνων, είναι σημαντικά εφόσον υπάρχει συνεργασία μεταξύ των σχετικών σώματων και φορέων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και στόχο του αναθεωρημένου προγράμματο δράση. Τέτοιου είδου σχέσει συνεργασία περιλαμβάνονται στου τρει βασικού οργανισμού στα θέματα τη θαλάσσια ασφάλεια, ιδίω στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή Frontex, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Ελέγχου της Αλίας ΕΦΚΑ και τον δικό μας. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να επιδιωχθούν οι στόχοι όπως δει. Οι στόχοι αυτοί και η σχέση ε, μεταξύ τους ήταν ένα από τα θέματα των αφηρημένων προγράμματος δράσης. Όμως θα πρέπει να οργανωθεί εντός των υπαρχουσών εντολών Πρέπει οι σχέσει συνεργασία να γίνουν ευφιέστερε, αποτελεσματικότερε και εν τέλει να προάγουν την καλύτερη δαπάνη των δημόσιων κονδυλίων, φεύγοντα τι επαναλήψει. Πριν ολοκληρώσω και κοιτάζοντα την ευρύτερη εικόνα, να πω ότι η ουσιαστική αξιοσημείωτη πρόοδο έχει επιτελεστεί σε ό,τι αφορά τι θαλάσσιε δυνατότητε, την έρευνα εντό των πρωτοβουλειών ασφάλεια και άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δεσμεύσει των κρατών μελών στην ΚΕΠΑ και τα πρώτα έργα, ε, προγράμματα ή επιχειρήσει ΚΕΠΑ εμέσω ή αμέσω έχουν σχέση με την υλοποίηση αυτού του προγράμματο δράση, όπω η παρακολούθηση στη θάλασσα, η προστασία των λιμένων, η θετική κινητικότητα. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με το υψηλό δυναμικό που προσφέρει η υλοποίηση του Ταμείου για την άμυνα. Το πρόγραμμα Οκεανή 2020 είναι πολύ σημαντικό για το πώς μπορούμε να ε, συνεργαστούμε σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ξεκίνησε πριν τον Αύγουστο και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό το μεγαλύτερο από τα τρία προγράμματα που επελέγησαν από τον διαγωνισμό το 2017 για την έρευνα στην άμυνα και ανοίγει το δρόμο για τέτοια ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα χρηματοδοτούνται από το Αμυντικό Ταμείο. Η υλοποίηση των αθεωρημένων προγραμματών δράση θα προωθήσει την θαλάσσια διάσταση σε όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε και εδώ θα πρέπει ο οργανισμό μα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να ολοκληρώσω, να τονίσω ότι η διαρκή δέσμευση των 100 μελών για την υλοποίηση αυτού του προγράμματο δράση και η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οργανισμού μας, καθώς και όλων των ε, οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγάλη σημασία. Όπως είπα στο παρελθόν, το επίπεδο συνεργασία μας με την ΕΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω για τα θέματα της θάλασσας, θα ωφελήσουν τα κράτη-μέλη και θα πρέπει όλα αυτά να θεωρηθούν αποτύπωμα για το μέλλον. Και γι' αυτό εκφράζω και τι ευχαριστίε μου, όλο ιδιαίτερα προ τη Βουλγαρική Προεδρία, για την ε, αφοσίωσή τη και τον ηγετικό ρόλο που ανέλαβε για να προωθηθούν τα θέματα αυτά. Παρόμοιες δεσμεύσει και τέτοια βούληση χρειάζεται και από τι επερχόμενε Προεδρίε για να έχουμε ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσω εγώ και μετά θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είμαι από παράκτια περιοχή, αλλά έχω σπουδάσει και το, την εξωτερική διεθνή ναυτιλία, το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ε, προς την Βουλγαρική Προεδρία που ασχολείται με το θέμα αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που εξετάζουμε το θέμα αυτό ως ΕΝΤΕ. Είχαμε μια θαυμάσια έκθεση από τον κύριο Πάσκου για τη Μαύρη Θάλασσα και εστιάζοντας κυρίως στα θέματα ασφάλειας της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Ήταν ε, ένα από τα κύρια θέματα που μας ε, απασχόλησαν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Επίσης, τουλάχιστον δύο φορές ε, ασχοληθήκαμε με την ασφάλεια της Βαλτικής. Και η ΑΦΕΤ και εμείς εδώ ως ΣΕΝΤΕ ασχολούμεθα με την ασφάλεια της Αρκτικής. Επίσης μας ενδιαφέρει λογικά το κέρας της Αφρικής. Που απασχολεί ιδιαίτερα και την EU Οπότε μια ερώτηση προς την ε, Προεδρία και τον ε, πρέσβη κύριο Χερτσίνσκι. Πώς εκτιμάτε τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit για το θέμα αυτό, για τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου για την ε, ανάπτυξη της ε, θαλάσσιας ε, ασφάλειας ήταν καθοριστική γιατί η χώρα αυτή είναι και μεγάλη και έχει και μεγάλη πείρα στα θέματα ελεύθερης ναυσιπλοείας. Επισκεφθήκαμε πέρυσι την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορες τακτικές μας συνεδριάσεις συζητήσαμε τα θέματα της ελευθερία της ναυσιπλοεία στην νότια θάλασσα της Κίνας και στην ανατολική Κινέζικη θάλασσα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα στα στενά μεταξύ Κίνας και Ταϊουάν. Και όλο και αυξάνονται, αυξάνεται η παρουσία στρατευμάτων στην περιοχή αυτή και επίσης ε, αυξάνεται και η παρουσία στρατευμάτων στην Ακτική. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γενικότερα στη Βαλτική. Στο Καλίνιγκραντ ε, περισσότερα στρατεύματα. Έχει ε, οικοδομήσει νέες εγκαταστάσεις εκεί η Ρωσία. Και η ίδια κατάσταση και στην Μαύρη Θάλασσα και η θάλασσα Αζόφ ιδιαίτερα θα μας απασχολήσει σε κάποια από τις προσεχείς συνεδριάσεις μας στη ΣΕΝΤΕ γιατί η κατάσταση σε αυτή την περιοχή όπως σωστά αναφέρθηκε στη Χερσόνησο του Κέρτς υπάρχουν ε, περισσότερα στρατεύματα αλλά όχι μόνο εκεί θα ήθελα τη γνώμη σας επ' Θα το συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γιατί και στην Αρκτική υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις αλλά ανησυχούμε για την κλιματική αλλαγή στην Αρκτική δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η δυνατότητα ναυσιπλοείας άρα θα υπάρχει και περισσότερος ανταγωνισμός και ίσως να αναπτυχθούν ακριβώς εκεί και ε, στρατιωτικές αντιπαραθέσεις και στην Μαύρη Θάλασσα. Ο κύριος Γκάλα και μετά η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Πολύ ενδιαφέρον ε, το πρόγραμμα δράσης και η εφαρμογή του ούτω ώστε τη στρατηγική αυτή να γίνει πραγματικότητα. Αλλά όπως είπατε αντιμετωπίζουμε πολλές και διαφορετικές προκλήσεις σε διάφορες περιοχές. Οπότε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Ντομέκ, αναφερθήκατε στην στρατιωτική κινητικότητα που είναι πρόγραμμα του project, του είναι πρόγραμμα του PESCO, συγγνώμη. Υποθέτω ότι στη θάλασσα είναι μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με τους δρόμους και τις ισοδομικές γραμμές που δεν είναι καθόλου προσαρμοσμένοι στις ανάγκες μας. Στη θάλασσα, άμα λειτουργούν οι μηχανές σου, μπορείς να κινηθείς. Υπάρχουν και συνδυασμένες μεταφορές ε, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες. Στην Ανατολική Γερμανία είχαν δημιουργήσει δυνατότητες συνδυασμού εγκαταστάσεων στην Ανατολική Γερμανία με εγκαταστάσεις στην ε, τότε Σοβιετική Λιθουανία από το Μούκραν στο Κλάιπεντα. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Θα μπορούσαμε ίσως να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς για στρατιωτικούς σκοπούς, δηλαδή συνδυασμένες και θαλάσσιες μεταφορές για να αυξήσουμε την ε, κινητικότητα των ε, στρατευμάτων μας. Για να υπάρξει κοινή οικοδόμηση δυναμικού, είπατε, και περιφερειακές ε, αντιδράσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις. Αναφερθήκατε σε περιοχές εκτός Ένωσης. Ο κόλπος της Γουινέας, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, έχετε σχέδια Εξετάζετε τις περιοχές όπου έχουμε φαινόμενα πειρατείας που απειλούν τις ε, θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Εδώ ε, στον τρίτο όροφο έχουμε την ισομερή συνέλευση ΑΚΕΟΚ όπου συζητάμε θέματα ασφάλειας της Αφρικής. Εφόσον λέμε ότι θέλουμε να είμαστε σε θέση να συμμετάσχουμε σε αποστολές CSDP, θα μπορούσαμε μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης των δυνατοτήτων ασφαλείας ή κάτι παρόμοιο και μέσω της συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες να αντιμετωπίσουμε κρίσεις σε αυτές τις περιοχές. Να βοηθήσουμε δηλαδή τις χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν οι ίδιες αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί αυτές οι χώρες στην Αφρική πρέπει να είναι κυρίως υπεύθυνε για αυτά που γίνονται στις ακτές τους για την καταπολέμηση της πειρατείας. Υπάρχουν ιδέες γι' αυτό. για να βελτιωθούν οι δυνατότητες σε μακρινές περιοχές να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Επίσης, πρέπει να διευρυνθεί ο μηχανισμός ε, Αθηνά. Ξέρουμε ότι η Πορτογαλία και η Ελλάδα για παράδειγμα έχουν ε, μεγάλο πολεμικό ναυτικό γιατί δεν μπορούν να συμβάλλουν λόγω του κόστους ε, χρήσης του ναυτικού τους. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θέμα μέσω του μηχανισμού Αθηνά της, του καταμερισμού του κόστους για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε διάφορα πολεμικά ναυτικά εάν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και ενημερώσεις. Αυτά που ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη αναφερθεί. Όπως για παράδειγμα αυτό που είπε η Πρόεδρος, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε για την κατάσταση εκεί. Ανάπτυξη συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σε συνδυασμό με, το, με τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ. Θα με ενδιαφέραν αυτά. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα. Και όπως είπαμε συζητώντας προηγουμένως την έκθεση Πάσχου. από την προηγούμενη εργασία στο ιατρικό τομέα και για αυτή την περιφερειοποίηση της προσπάθειάς μας, φυσικά η Δυτική ε, Μεσόγειος μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Τι επιτυχίες θεωρείτε ότι είχαμε σε αυτή την εντολή παρεμπόδισης που δόθηκε στη Σοφία. και πώς θα συνεχιστούν στα πλαίσια του προγράμματος δράσης που συζητάμε. Ένα άλλο θέμα. Η, τα υποθαλάσσια καλώδια. Κύριε Φρύς, αναφερθήκατε σε αυτό. Τα καλώδια αυτά είναι ζωτική σημασία για τις τηλεπικοινωνίες μας. τι απειλέ μπορεί να υπάρχουν για αυτά τα καλώδια και πώς θα τα προστατεύσουμε. Και τελειώνω. Κύριε Ντομέκ, είπατε ότι γίνεται έρευνα λόγω της χρηματοδότησης που δίνει η Ένωση μέσω του ορίζοντα 2020 για τα προϊόντα διπλής χρήσης και με διάφορα πολιτικά προγράμματα. Πού θα πρέπει να εστιάσει στο μέλλον η έρευνα για τα θέματα αυτά. Και τέλος, με χαρά άκουσα όλους τους ομιλητές να λένε ότι υπάρχει συντονισμός, οριζόντια συνεργασία, ότι είναι αναγκαία και ότι θεωρείται ότι βελτιώνεται. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Για παράδειγμα, για θέματα ασφάλειας και εσωτερικών. Πώς θα αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, τους δορυφόρους μας. Πώς θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, νομίζω ότι κλείνουμε έτσι τον καταλότρο μιλητών. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Ε, θέλω όμως να προσθέσω κάτι. Σε όλες τις ε, λεκάνες τις οποίες αναφέραμε, Μεσόγειο, Βαλτική θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ε, Αρκτικός, Οκεανός κλπ. Η, ε, η παρουσία μας συνδέεται και με ενεργειακά προγράμματα και σχέδια εξαιρετικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η ναυσιπλοεία εκεί είτε περιορίζεται είτε απειλείται και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ενισχύσουμε την ασφάλεια ασφάλεια, μιλάμε για ε, τρομοκρατικές απειλές, κυβερνοασφάλεια κλπ. Ε, η κυρία Καρατζόβα σχολίασε ορισμένα από αυτά, ορισμένες από αυτές τις απειλές. Υπάρχει μια περιφερειακή τοπική έμφαση για κάθε μία από αυτές τις ε, λεκάνες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρατζόβα, τον ε, πρέσβη κύριο και τον ε, πρέσβη κύριο Ντομέκ επίσης. Καταρχήν κύριε Καρατζόβα. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ που μας ε, ε, υπογραμμίζετε το θέμα της Μαύρης Θάλασσας. Για μας είναι και θέμα εθνικής προτεραιότητας. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στην αρχική μου παρουσίαση. Παρ' όλα αυτά είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας έτσι ώστε το πρόγραμμα δράσης να είναι ισόρροπο γεωγραφικά. Στη Μαύρη Θάλασσα προβλέπουμε συγκεκριμένες ε, δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις σχετικά με τη θάλασσα ασφάλεια. Θα στηρίξουμε συνέργειες ε, για από την, ε, μέσω της ε, ε πρωτοβουλίας για την περιοχή. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει πολύ σημαντική γεωπολιτικά, αλλά για τους κακούς λόγους, για όχι για τους σωστούς λόγους, ε, στρατιωτικοποιείται μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, παρά, παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 από τη Ρωσία, η συνεργασία στην περιοχή αυτή για θέματα ασφάλειας είναι πολύ περιορισμένη για να μην πω έχει παγώσει Έχουμε μόνο το έγγραφο για τα μέτρα ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ενώ οι, όλες οι άλλες πρωτοβουλίες όπως οι, των τεσσάρων της Μαύρης έχουν παγώσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες να συνεργαστούμε σε άλλες σε άλλους τομείς όπως παράνομες δραστηριότητες ε, η προστασία των ενεργειακών υποδομών, το περιβάλλον, τις μεταφορές. Μαζί με τη Ρουμανία ε, θα προσπαθήσουμε να ε, εστιάσουμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες ε, μετά τη συνάντηση των Μπουργκά στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Μέχρι το τέλος του μήνα θα συναντούν οι Υπουργοί Εξωτερικών μας. Επίσης, μας ικανοποιεί η έμφαση που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Μαύρη Θάλασσα στην έκθεση που εγκρίνατε αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα αυτόνομα. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ και καιρό το επισημαίνουμε. Παρόλο ότι υφίσταται από το 2007 η διαδικασία για την, πρωτο... για την πρωτοβουλία για τη συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα, και υπάρχει και διασυνοριακή συνεργασία στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, έχουμε πάρα πολλά που υπολείπονται. Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, ειδικά σε αυτήν την περιοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για προφανείς λόγους. Τα σχέδια της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας επίσης σχετίζονται και με τη Μαύρη Θάλασσα. Ε, τα συστήματα, αυτόνομα συστήματα ε, θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς επίσης και τα συστήματα παρακολούθησης θάλασσα πρέπει επίσης να ενισχυθούν. Μετά, συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Πράγματι, αναμφίβολα θα χρειαστεί να ενισχυθεί. όπως και μέσω της συνεργασίας μας με τον ΝΑΤΟ. Όμως ε, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μετά το Brexit για να διαπραγματευτούμε μια μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτό το θέμα. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να καθορίσουμε λεπτομέρειες για την μελλοντική μας σχέση αυτή τη στιγμή διεξάγουν διαπραγματεύσει ακόμα για τον Brexit. Ε, υπάρχουν ήδη βέβαια θέματα για την ε, επιχείρηση Αταλάντα και την, ε, ε τον ορισμό διοικητή ε, θα τα εξετάσουμε σύντομα. Ο ε, κ. Φρύς σε ό,τι αφορά τον αρκτικό, την αρκτική ζώνη, με το λιώσιμο των πάγων, πράγματι, είναι πιθανό να ανοίξουν καινούριε δύο μεταφορικές ε, μέσω του Αρκτικού ωκεανού. Μεταφορές που θα έχουν σχέση και με τον τουρισμό αλλά και με τα εμπορεύματα. Ε, και ενδεχομένως μάλιστα και μεταξύ ε, διαφορετικών υπήρων, δηλαδή από την Αμερική προς την Ευρασία κλπ. Το, οι αλλαγέ του, στο κλίμα ε, προφανώς ε, θα επηρεάσουν και την οικονομία. Είναι βέβαια ε, λιγότερο από τι επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία αυτή τη στιγμή, λιγότερο από ό,τι περιμέναμε πριν από μερικά χρόνια. Σίγουρα όμως θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην ασφάλεια. Ο Αρκτικός Ωκεανός αυτή τη στιγμή διακυβερνάται με ένα σχετικά συνενετικό τρόπο μέσω του Συμβουλίου του Αρκτικού Ωκεανού η ομάδα των χωρών που το απαρτίζουν φαίνεται να καταλήγει σε πρακτικά και εφαρμόσιμα συμπεράσματα και για την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρήτρια στο Συμβούλιο του Αρκτικού. Τα δύο, υπάρχουν όμως δύο κράτη-μέλη μας που είναι μέλη. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο από την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να σχολιάσει θέματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα σχολιάσω το θέμα της στρατιωτικοποίησης, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό που θέλουμε είναι να ε, αναπτύξουμε ικανότητες σε θέματα ασφάλειας και άμυνας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Στη Μαύρη Θάλασσα θα συμφωνήσω με την κυρία Καρατζόβα. Η περιοχή αυτή είναι κρίσιμη, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τούτου λεχθέντος είναι δυνατόν, κατά την άποψή μας, να αντιμετωπίσουμε από καινού θέματα ασφάλεια στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα μια κλειστό χώρο ε, που ε, και επιβαρύνονται όλοι οι γείτονε, όταν, για παράδειγμα, συλλαμβάνει η χώρα υπεραλίευση ή η μόλυνση των υδάτων κλπ. Οι, οι, οι, υπουργοί, οι των χωρών γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα το Μάιο κατέληξαν σε μια, ενέκριναν μια δήλωση που περιλαμβάνει θέματα στα οποία είναι δυνατόν να γίνει συνεργασία. και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδου δραστηριότητε, προφανώ κυρίω προ συμφέρον των δικών μα μελών. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Σοφία και την Μεσόγειο, εγώ θέλω να πω απλώ ότι η η συνεργασία ανάμεσα στις τρεις υπηρεσίες που σχετίζονται και η ανταλλαγή πληροφοριών, οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί σίγουρα συνεισφέρουν στην ε, επιχείρηση Σοφία. Για τα υποθαλάσσια καλώδια ε, περιλαμβάνονται στις ε, κύβερνοαπειλές στο κείμενο. Θα πρέπει πρώτον να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν αυτό πόσο κινδυνεύουν οι υποδομές αυτές. Θα πρέπει να, αξιολογηθεί, να αξιολογηθούν το αν χρειάζονται προληπτικά μέτρα και ποια μέτρα. Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό το ζήτημα και υπάρχει λόγο να γίνει, είναι σοβαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σερτίνσκι, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κάποιες από αυτές δεν είναι εύκολο να απαντηθούν, αλλά θα αποπειραθώ. Μία προς μία. Ξεκινώντας με το τι αντίκτυπο θα έχει το Brexit. Ιδίως στην επιχείρησή μας Αταλάντα είναι σαφέ ότι η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην όλη επιχείρηση εδώ και χρόνια ήταν καθοριστική σημασία και δεν είναι τυχαίο που το Γενικό Επιτελείο βρίσκεται στο Northmouth, ε, κοντά στο Λονδίνο. Βεβαίω δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω τα ξέρετε. Και όπω ακριβώ τα ξέρετε, συζητήσει για το μέλλον το στατικίου μας, του γενικού μας επιτελείου, είναι κάτι που ε, πολλά κρατημέλη το ε, θέλουν και διαγωνίζονται μεταξύ τους αυτή τη στιγμή. και το πρώτο πάρει από το Northwood. Northwood. Όμως ε, η θετική εμπειρία από την επιχείρηση αυτή είναι κάτι που θέλουμε να συνεχιστεί. Από το 2012 Υπάρχει σοβαρή μείωση στις επιθέσεις πειρατών από το 2008 έως 2011 υπήρχαν 571 ε, ε, επιθέσεις, 136 ήταν από πειρατές, ενώ ε, από το 2013 είχαμε 18 επιθέσεις συνολικά και μόνο δύο από αυτές ήταν από πειρατές. Άρα σαφώς και υπάρχει διαφορά. Τι θέλουμε να κάνουμε, να διαφυλάξουμε ακριβώς όσα καταφέραμε στον αγώνα κατά της πειρατείας στο κέρας της Αφρικής. Καθώς και τους μηχανισμούς και τις σχέσεις συνεργασίας που ε, επιτυχώς δημιουργήθηκαν όπως ο μηχανισμός SAID για την ευαισθητοποίηση, το κέντρο για το επιχειρησιακό κέντρο για το Κέρας της Αφρικής ΚΟΑ, καθώς και το κέντρο εκτοφυλακή στην ακτή τη Ομαλία, για τη μελλοντική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είπε και η πρέσβυρα Καρατζόβα. είναι μέρος της ενεξελίξης συζήτησης αυτό και ίσως να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέψει καλύτερη συνεργασία και συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Και βεβαίως εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις για τα άλλα θέματα. Για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της ε, Μαύρης Θάλασσας, του Αυξήνου Πόντου δηλαδή και του Αρκτικού Ωκεανού, ε, και της Βαλτικής θα υπάρξουν δύο δυνατότητες οι αρχηγοί μας να συζητήσουν τις δόλιες δραστηριότητες της Ρωσίας τις ερχόμενες εβδομάδες. Πρώτα απ' όλα, στη σύνοδο του Σέλσπερι, μάλλον με την επίθεση του Σέλσπερι, όπως ξέρετε το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, την Άνοιξη ανέθεσε και στην υπατή εκπρόσωπο και στην Επιτροπή να ενημερώσουν για την ε, συνέχεια που δόθηκε στις επιθέσεις του Σέρσπερι και η έκθεση αυτή εγκρίθηκε μόλις τις 13 Ιουνίου πριν από λίγες μέρες. Πολύ ξεκάθαρα περιγράφει τι απόκριση θα πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υβριδικά κυβερνοεγκλήματα ή εγκλήματα μυστικών πληροφοριών. Ε, δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων την ερχόμενη εβδομάδα είναι τι να γίνει με τις οικονομικές, τι πρέπει να γίνει με τις οικονομικές κυρώσεις ε, κατά της Ρωσίας. Και εδώ υπήρχε ένα εξάμεινο περιθώριο για αποφάσεις. Βεβαίω δεν μπορούμε να προδικάσουμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση, αλλά μπορούμε να φανταστούμε κάποια μετακύληση καθώς αυτά τα οικονομικά μέτρα ε, εξαρτώνται και από την όλη κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία και τη διαδικασία του Μίνσκ. Εάν δεν υπάρξει καμία πρόοδο στη υλοποίηση της διαδικασίας του Μίνσκ, δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξουμε τη στάση μας. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα που θα συζητηθούν Τώρα για την CBST, την Αφρική, το κοινό κόστος και την επιχείρηση Αθηνά. Είναι πολύ εύστοχα όλα αυτά, επειδή ξεκίνησε η συζήτηση για το νέο εργαλείο, το λεγόμενο διευκόλυνση για την ειρήνη. Κάτι που άρχισε να εξετάζεται από τα κάτι μέλη πριν από μια-δυο μέρε. Βεβαίω έχουμε και το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο το 2020, αλλά δύο από τα τρία στοιχεία της διευκόλυνσης για την ειρήνη είναι ακριβώς να συνδυαστεί το κοινό κόστος και να αυξηθεί σημαντικά, δηλαδή να υπάρξει ταχύτερη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την εκδίπλωση και την αποστολή στρατευμάτων και συγκεκριμένα να ενισχυθεί η οικοδόμηση δυνατοτήτων σε τρίτες χώρες. Όχι με έμφαση μόνο στην Αφρική, αλλά αυτή η δυνατότητα να προβλέπεται διεθνώς. Αυτό που κάνουμε βεβαίως ως τώρα, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, ήταν και παραμένει προτεραιότης. για την επιχείρηση Σοφία η ε, στόχος της όπως ξέρετε αρχικά ήταν να ε, χτυπήσει, να πλήξει το business model για να το πω έτσι, το επιχειρησιακό μοντέλο των ε, λαθρεμπόρων ανθρώπων. Πολύ γρήγορα πέρασε στο να διασώζει ζωές στη θάλασσα η όλη επιχείρηση. Βεβαίω δεν έχω μαζί μου τα σχετικά στοιχεία, όμω υπήρξε ένα σημαντικό αριθμό λάθρεμπόρων που συνελήφθησαν και σκαφών που καταστράφηκαν. Διαλύθηκαν. Ε, προστέθηκαν και άλλες αρμοδιότητες στην επιχείρηση Σοφία με την πάραδο του χρόνου και ένα ε, από αυτά που προσθέθηκαν ας πούμε, και πρέπει να αναφέρω είναι η εκπαίδευση της Λιβικής Ακτοφυλακής. Είναι εξελίξη διαδικασία και δύσκολη, όμως έχει πολλές προοπτικές να αλλάξει την κατάσταση. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και εσείς τώρα, πρέσβη ναι, ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Για αυτό που ο κύριος Γκάλερ για τη σερβική ασφάλεια. Όταν μιλάμε για τη θάλασσα, δεν μιλάμε μόνο για τις υποδομές, αλλά και τη διασύνδεση ξηράς και θάλασσας. Στον τομέα λοιπόν της ταχυδικής κινητικότητας, ιδίω για τη θάλασσα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με τεχνολογίες που σχετίζονται και με συστήματα μη επανδρομένα για το μέλλον της θάλασσας. Κάτι που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Για την ερώτηση της κυρίας Μοντή για την έρευνα, βασική έμφαση στην όλη προσπάθεια δίνεται με την Ευρωπαϊκή Ιστιτωτική Ατζέντα, την Ατζέντα μάλλον της Ειδικής Έρευνας, που εκδώσαμε σε συνεργασία με την ΕΓΕΔ πέρσι στις 18 Δεκεμβρίου. Και εδώ αναφέρονται οι τομείς που θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε διατομεακά. Μπορώ να σας διαβάσω μερικούς από τους τομείς. Ε, ε παρακολούθηση, διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων, αυτόνομα συστήματα έρευνες και πλατφόρμες πολλαπλής χρήσης. Όπως είπατε για τη διατομιακή προσέγγιση που ζητά και το πρόγραμμα δράσης, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ε, ολοκληρωμένο. Είναι μια ενεξελίξη διαδικασία και όπως είπα, Υπάρχουν τομείς που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε τους διαχωρισμούς μας, τα θεωρητικά πράγματα και ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Εδώ έχουμε πολλές διαφορετικές ομάδες και που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία. Ένα παράδειγμα, ένα πετυχές παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν. Δύο παραδείγματα. Διεξαγάγαμε ένα τεστ για τη χρήση κάποιων συστημάτων στην Μεσόγειο της Μάρσουρ εκεί είδαν κατά πόσο ήταν ε, αποτελεσματική η χρήση και από τον οργανισμό μας και από τη Μάρσουρ και ένας άλλος χώρος που βλέπουμε ε, συνδυασμό είναι τα σεμινάρια εκπαίδευσης για την ε, διαχείριση της κρίσης των μεταναστών. Το προσωπικό μας δεν είναι αναγκαστικά εκπαιδευμένο σχετικά, όμως ταυτόχρονα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τους συνοριοφύλακες και τους ακτοφύλακες, όχι μόνο τους εθνικούς, αλλά και τις Frontex. Έτσι λοιπόν έγινε ο πρώτος γύρος εκπαίδευσης πρόσφατα και βλέπουμε με τη Frontex πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τα δορυφορικά, η θέση των 100 μελών και του οργανισμού για όλα τα θέματα που αφορούν το διάστημα και τα διαστημικά προγράμματα είναι στον βαθμό που γίνεται από την αρχή και δεν μιλάω για αυτά που ήδη λειτουργούν πλήρως όπω ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος οι στρατιωτικές απαιτήσει να ενσωματωθούν από την αρχή ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και σκοπούς στρατιωτικούς και πολιτικούς. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως δημοσιεύτηκε πέρσι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, πρέσβη Ντεμέκ, νομίζω ότι με αυτά ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για την ε, στρατηγική της θαλάσσιας ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει ε, επικαιροποιηθεί και τις αλλαγές στο πρόγραμμα δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ χειροκροτήστε μαζί μου τους εξαιρετικούς μας αποστοιχημένους. Thank you. Uh, ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι ξεκινάμε στις 2.30 ακριβώς μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας.